Κύριε στην έναρξη τη ε, σημερινή μα ε, απογευματινή συνεδρίαση, η βραδινή συνεδρίαση. και καλωσορίζω βέβαια και την Επιτροπή Προπολογισμών η οποία μπορεί να συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίασή μα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο και του δημοσιονομικούς ε, κανόνε. καταρχήν έχουμε την ημερήσια διάταξή μα μπροστά μα, την εγκρίνουμε λοιπόν. Από εκεί και μετά στο δεύτερο σημείο έχουμε τα cont news. Γνωρίζετε τι συμβαίνει εκεί, γνωρίζετε ότι υπάρχει και web streaming, ολόκληρο ο τύπο ε, μα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα. Ε, και μετά βέβαια έχουμε και ένα πολύ σημαντικό σήμερα, ε, σήμερα σε ό,τι αφορά την Guardia τη Φινάνσα και τις ταλικές αρχές και χαίρομαι που θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά το σημείο 3, εγώ ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι αρμόδια και θα ήθελα να ζητήσω από, ε, συγγνώμη από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για το γεγονό ότι ο συνάδελφο δεν παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Θα ήθελα να σα ενημερώσω σε ό,τι αφορά τι τελευταίε δύο συνεδριάσει του τριμερίου διαλόγου στι 7 και 11 Νοεμβρίου ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση Omnibus ε, και συζητήσαμε τα άρθρα 176 έως 228 των δημοσιονομικών κανόνων και φτάσαμε σε μια προσωρινή συμφωνία σε σχέση με τα εξή άρθρα το 79 καταρχήν τα usual cost accounting practices, το 80 ε, τα σημεία που ε, εγκρίνονται για ενισχύσεις, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της εθελοντικής εργασίας. Υπάρχει το άρθρο 181 σε σχέση με τις ε, συνδεδεμένες οντότητες, affiliated entities, και εδώ φτάσαμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά και το 182 και το 185 και 186 σε ό,τι αφορά τις ε, επιχορηγήσεις ε, και την απαγόρευση της ε, αθρηστικής τους προσμέτρησης αλλά και της αναδρομικής χρηματοδότησης. Στα 187 και 188 συζητήσαμε τις, τους προκηρύξεις και 198 συζητήσαμε τα κριτήρια επιλογής και της επιλογής των πλειοδοτών στο άρθρο 200 συζητήσαμε επιμέρους ζητήματα σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις για τα πράγματα γιατί γνωρίζετε πως πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, ε, για το οποίο δηλαδή υπάρχει ε, ένα εφάπαξε πλέον ε, ποσό που διαθέτει η ε, ένωση. Ε, στο άρθρο 203 συζητήσαμε σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, ενώ το 210 συζητήσαμε με τα όργανα ε, διοικητικού χαρακτήρα. Άρθρα 211 και 212 αναφερθήκαμε εδώ στις εγγυήσεις του προπολογισμού και συζητήσαμε στα άρθρα 214 και έως 226 της πολιτικής ομάδας ενώ υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη ε, και ένα σημαντικό σημείο ε, που παραμένει κρεμές στα 215 έως 219. Σε ό,τι αφορά τους εξπόστ ελέγχους και τα καταποκοπή ποσά, τα λάμψαμς, δεν φτάσαμε ακόμα σε συμφωνία αλλά ε, και τα ποσοστά σε ό,τι αφορά την εθελοντική εργασία, τους κανόνες διαφάνειας, τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, και σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε μεγάλες διαφορές απόψεων με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το καινούριο ταμείο αλλά και το ζήτημα των καταπιστηματικών ταμείων, των trust funds και τις σχετικές υποχρεώσεις και γι' αυτό έχουν προβλεφθεί και περαιτέρω συνεδριάσεις τριμερούς ε, διαλόγου, πέντε συνεδριάσεις, 20 Νοεμβρίου, 27 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου, 6 Δεκεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου. Πέντε λοιπόν συνολικά συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου. Ε, λάβαμε ακόμα απόψη μα ότι ο τιμερή διάλογο στι διάφορε επιμέρου επιτροπέ έχει ολοκληρωθεί και γνωρίζουμε πω το αγροτικό τμήμα, που βέβαια δεν αφορά άμεσα του δημοσιονομικού κανόνε, θεωρήσαμε πω δεν θα περιληφθεί στο πλαίσιο τη συζήτηση τη πρόταση Όμνιμπου, έτσι ώστε να επιτύχουμε πρόοδο και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου και στο επίπεδο του Συμβουλίου. Δηλαδή αυτή είναι η πρόταση να ασχοληθούμε ξεχωριστά με το αγροτικό τμήμα έτσι ώστε ε, τα υπόλοιπα σημεία μπορούσαν να ισχύσουν από το ε, Ιανουάριο. Ε, τα ζητήματα των τραν ε, δεν μπορούμε να τα εξαιρέσουμε ούτε τα ζητήματα της ΡΕΚΙ γιατί υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προπολογισμού και κατά συνέπεια σχετικέ αρμοδιότητε αυτή τη ΡΕΚΙ. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση από την δική μου πλευρά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερωτήματα. Ο συνάδελφο Χουμπίχη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, παρουσίαση. Αυτό που θα με ενδιαφέρε εμένα σε αυτή τη φάση είναι το γεγονός ότι πολλά έργα όπως ε, το Ταμείο για την Αφρική υλοποιούνται αυτή την ε, περίοδο, αλλά θα πρέπει να προσανατολιστούμε ταυτόχρονα και στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και υπάρχει το, το 2 για την για την ε, γεωργικό τομέα, ενώ το SD7 σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα project τα οποία εκτελούνται, αλλά εάν ένα έργο εκτελείται μεμονωμένο, τότε ε, συχνά η αρχιτεκτονική αλλά ταυτόχρονα και η συντήρηση για παράδειγμα ενός τέτοιου έργου δεν ε, συνδέονται μεταξύ τους, λαμβάνουν χώρα δηλαδή αυτόνομα. Δεν θα έπρεπε ε, να προβλέψουμε για παράδειγμα ε, ξεχωριστά έναν ε, διαγωνισμό σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μετά στο δεύτερο κομμάτι το κατασκευαστικό τομέα και μετά μία ακόμα προτήρηση σε ό,τι αφορά 30 ετή συντήρηση, για παράδειγμα, και διασφάλιση ότι θα λειτουργεί καλά μια εγκατάσταση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ε, έχω διαπιστώσει ότι στο παρελθόν αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ναι, μεν κατασκευαζόταν ε, για παράδειγμα μια εγκατάσταση, αλλά ταυτόχρονα μετά από λίγο καιρό πάβε να λειτουργεί. Οπότε οπουδήποτε εμεί προβλέπουμε κάτι τέτοιο, είτε πρόκειται για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, είτε πρόκειται για το γεωργικό τομέα, θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι ακριβώ θα λειτουργήσει σωστά και στο μέλλον. Οπότε ίσω θα πρέπει να ε, προβλέψουμε ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ναι, επί τη αρχή συμφωνώ μαζί σα, αλλά εξαρτάται κάθε φορά από το σε ποιο τομέα βρισκόμαστε και σε ποιο ταμείο αναφερόμαστε. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ξεχωριστά το κάθε ταμείο και βέβαια στο πλαίσιο του κοινού νου αν θέλετε να επιτύχουμε ακριβώς κάποιους ε, τέτοιους κανόνες. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να δούμε τι προβλέπεται στο ουσιαστικό δίκαιο. Και αυτό προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανόνες του προπολογισμού είναι το γεγονός ότι οι επενδύσεις αποτελούν διαφορετικό είδος απόφασης και μπήκουν σε μια διαφορετική διαδικασία προκήρυξης. Αλλά θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι γίνεται ξεχωριστό διαγωνισμό για, για τέτοιε επενδύσει. Δηλαδή, ένα διαγωνισμό για την κατασκευή και ένα άλλο διαγωνισμό σε ό,τι αφορά τη συντήρηση. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Αλλά ακριβώ επειδή είναι δυνατόν να γίνει ήδη κάτι τέτοιο, ίσω δεν κατάλαβα σωστά τον συνάδελφο Γουίμπη γιατί προτείνει να αλλάξει κάτι ήδη επιτρέπεται αυτό. Αλλά, εν πάση ίσω θα μπορούσατε να συγκεκριμενοποιήσετε λίγο το έτοιμά σα για να ε, δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και υποστηρίζω εδώ, ε, συγγνώμη, καλωσορίζω εδώ και τον ε, πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Προπολογισμών. Αναφέρθηκα στο, στα σημεία στα οποία καταφέραμε να συμφωνήσουμε και σε εκείνα που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε και το γεγονό ότι θα λάβουν ακόμα πέντε συναντήσει στο πλαίσιο του τριμερού σε διαλόγου. Αλλά βλέπω πω ο συνάδελφο Τσέλα έχει θέσει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, κατά τη δική μου άποψη και καθώ ε, έχω ασχοληθεί στο παρελθόν και με την εφαρμογή των τελών τη Ένωση, έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι ε, δημιουργεί κάποια κίνητρα η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση μέσω τη χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση συγκεκριμένων επενδύσεων αλλά η συνέχεια που δίνεται σε αυτές τις επενδύσεις είναι κάτι το οποίο επαφίεται πλέον στον δικαιούχο ε, και δεν χρηματοδοτείται πλέον από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και αυτό βέβαια οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ανέφερε σωστά και ο συνάδελφος Παύλο να προκύπτουν ζητήματα, όπως έχω και εγώ διαπιστώσει σε μια σειρά από κράτη-μέλη. Δηλαδή επενδύσει οι οποίε υλοποιούνται, αλλά στη συνέχεια δεν λειτουργούν, γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει το κατάλληλο καταρτισμένο προσωπικό, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί τελικά πόροι. Οπότε έχουμε δει σε ορισμένε περιπτώσει, παρότι υπάρχει σωστή πρόθεση, το αποτέλεσμα να μην είναι εκείνο το οποίο επιθυμούσαμε. Την περασμένη, για παράδειγμα, εβδομάδα συναντήθηκα με διάφορου εκπροσώπου τη ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών από αφρικανικέ χώρε, στου οποίου είχαμε υποσχεθεί πριν από δύο χρόνια στη Βαλέτα ότι θα υπάρξουν τέτοιου είδου χρηματοδοτήσει επενδύσεων στην ε, Αφρική. Με ρώτησαν λοιπόν τώρα αυτοί οι εκπρόσωποι τη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών πότε θα ξεκινήσει αυτή η χρηματοδότηση των λόγω έργων. Γιατί δεν βλέπουν ακόμα να έχει λάβει χώρα κάτι απτό, κάτι ορατό. Ε, Στι ε, χώρε του. Ε, και εγώ βέβαια δεν ήμουν σε θέση να του δώσω μια απάντηση γιατί αυτού, αυτού του είδου οι επενδύσει δεν ευήκουν στον τομέα αρμοδιότητα το δικό μα. Προεδρο. Ναι, ίσω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε διμερώς λίγο αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή πω πραγματικά θα πρέπει να και σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των στόχων μα. Αλλά εάν ε, θέλουμε πραγματικά όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε, δηλαδή ζητήματα που αφορούν 6 και 10 χρόνια από τώρα, δεν θα καταλήξουμε πουθενά τελικά. Οπότε θα ήθελα σε αυτή τη φάση να ολοκληρώσουμε το σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη και να περάσουμε στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Οι δραστηριότητε δηλαδή κατά πόλεμη τη απάτη στην Ιταλία. Ε, και εδώ καλωσορίζω ε, θερμά τον Υπουργό Περόλα, ο οποίο είναι ο επικεφαλή της γραμματείας ενός ε, διυπουργικού συμβουλίου σε ό,τι αφορά εξωτερικές υποθέσεις και αναμένουμε εδώ και τον ε, διοικητή της Γκόρτα τη Finanza, τον κύριο Τόσκιν και ε, τον υποστράτηγο Φρανσέσκο Ατάρντι, ο οποίος επίσης για την Κόρτα di Finanza Ε, οπότε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βερόλα, σας καλωσορίζουμε θεμά και μπορείτε να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχάς ε, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για τη δυνατότητα που προσφέρατε στην Guardia di Finanza και στην ε, Ιταλική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης, την ΑΦΚΟΣ, να σας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Ιταλίας για τον τομέα αυτό. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, να σας διαβάσω και τους χαιρετισμού ε, του Υπουργού ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ε, του Σάντρο Γκότση, ο οποίος έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, ο οποίος δυστυχώς όμως χρειάστηκε να παραμένει στη Ρώμη, διότι προέκυψαν κάποιες πολιτικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να ταξιδέψει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς, να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές που είναι παρόντες, αλλά και την Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού για την ευκαιρία αυτή. Ξέρω ότι ο στρατηγός ε, Τόσκι και ο στρατηγός ε, Ατάρντι ε, μέχρι πριν από λίγο ε, ήταν ε, σε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Μου γνέφουν εδώ οι βοηθοί τους ότι όντως, αλλά είναι καθοδόν, είναι εδώ στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου και από στιγμή σε στιγμή θα καταφτάσουν. Επιτρέψτε μου λοιπόν κυρία Πρόεδρε να αφιερώσω εγώ κάποια λεπτά για να σας παρουσιάσω λίγο το περιεχόμενο αυτής της παρουσίασης και το πνεύμα βάσει του οποίου δραστηριοποιούνται οι Ιταλικές αρχές, η κυβέρνηση και η Guardia του Finance ε, για να παρουσιάσουν εδώ ε, στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο τις δραστηριότητες ε, στο συγκεκριμένο τομέα από πλευράς Ιταλίας. Σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα σας ε, παρουσιάσουμε καταρχάς ε, τις δραστηριότητες υπηρεσίες συντονισμού καταπολέμησης της απάτης, της Ιταλικής δηλαδή υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης. Δεν θα δείτε μόνο τις δραστηριότητες, αλλά και τις οργανωτικές αρχές, αν θέλετε, και ε, θα σας παρουσιάσουμε και αυτό το ε, έργο συνεργασίας ε, για την καταπολέμηση της απάτης. Νομίζω σας έχει ε, διανεμηθεί και αυτό το βιβλίο στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες ε, της υπόθεσης. Μετά θα δώσω το λόγο στο στρατηγό Ατάρντι, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής ε, του τμήματος της μονάδας που είναι αρμόδια για την πρόληψη της απάτης της βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Καταπολέμησης Απάτης της Ιταλίας. Εγώ θα περιοριστώ σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την εθνική στρατηγική. Όπως θα γνωρίζετε ίσως ε, εσείς στην Επιτροπή σας, η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία του προπολογισμού της Ένωσης είναι κοινή αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών. Είναι όμως πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές ε, να ε, συμμετέχουν ενεργά και πραγματικά να θεωρούν ότι είναι μεταξύ των καθηκόντων τους να καταπολεμούν την εθνική απάτη, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δραστηριότητες ε, οι οποίες γίνονται επιτόπου ε, να αντιμετωπίζονται επιτόπου διότι δεν είναι πολύ εύκολο από τις Βρυξέλλες, από το Στρασβούργο ή οι ευρωπαϊκές αρχές ε, να διώκουν υποθέσεις απάτης οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Χρειάζεται λοιπόν να διαθέτουμε εθνικές αρχές οι οποίες θα έχουν τα κατάλληλα κίνητρα αλλά θα, και την κατάλληλη δομή επιτόπου, αλλά θα πρέπει επίσης οι εθνικές αρχές να συνεργάζονται και μεταξύ τους εκφύσεως ε, ε, των εγκλημάτων ε, και των παράνομων δραστηριοτήτων που είναι εις βάρος του κοινοτικού προπολογισμού. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί πάρα πολύ ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να δοθούν ε, πολύ ισχυρά κίνητρα στις εθνικές αρχές και να τις προσανατολίσουμε προς αυτές τις δραστηριότητες. Ακόμα και σήμερα όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές ε, στο επίπεδο δέσμευσης ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Η κοινή δέσμευση λοιπόν θα πρέπει να είναι να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμει όλων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων για να ε, επιτύχουμε αυτό τον κοινό στόχο. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ιταλία και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα έχει ε, καταλήξει σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα με αυτό θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στον ε, στρατηγό Ατάρτη, ο οποίος θα σας παρουσιάσει αναλυτικά αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ θα περιοριστώ σε ε, ένα αποτέλεσμα, το οποίο ίσως ε, καταδεικνύει και τον αντίκτυπο που έχει όλη αυτή η δουλειά. Η δραστική μείωση τα τελευταία δύο χρόνια των εισαγωγών που αφορούν περιπτώσεις απάτης ε, λόγω παρατυπίας που διαπιστωνόταν στην Ιταλία. Από το 62% που είχαμε το 2015 μέχρι σήμερα ο αριθμός ε, ε, αυτών των παρατυπιών μειώθηκε, συγγνώμη, ο αριθμός μειώθηκε κατά 62% από το 2015 και από εκεί και πέρα ο κύριος Ατάντη θα σας παρουσιάσει το ποσοστό μείωσης του περιθωρίου σφάλματος που είναι ο όρος που χρησιμοποιείται επίσημα για αυτά τα σφάλματα και τον πολύ καλό τρόπο με τον οποίο ε, κάποια θέματα και κάποιες συστάσεις της Όλαφ. Ε, θα ήθελα με αυτόν τον τρόπο να... Ε, ευχαριστήσω και δημοσίως ε, το, η μονάδα αυτή που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ εντάχει είναι η Ευρωπαϊκή Όθηση. Ο στρατηγός Ατάρδη και ο στρατηγός Τάοσκι ίσω θα μπορούσαν να σας πούν κάποια περισσότερα για το θέμα, διότι είναι πλέον οι δήμονες σε σχέση με μένα αλλά να σας πω επίσης ότι η μονάδα μας δραστηριοποιήθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενθαρρύνει να υπάρξει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Και αυτό έγινε προτείνοντας ε, συνεχώς ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις ευρωπαϊκές δομές ε, μια πιο ισχυρή διοικητική συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ εθνικών αρχών και αυτό έγινε και μέσω και ε, κάποιων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που πρότεινε αυτόνομα. Ο στρατηγός Ατάρντι ίσως θα μπορέσει να σας πει κάποια πράγματα παραπάνω και να επεκταθεί λίγο περαιτέρω. Πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη από ε, εθνικές αρχές των κρατών μελών ε, της Ένωσης και χωρών που έχουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης, όχι μόνο υποψήφιες χώρες για προσχώρηση και αυτές οι δραστηριότητες τελικά μεταφράστηκαν σε μία σειρά από εταιρικέ σχέσεις, ε, συμπράξεις ε, με άλλους ε, μονάδες καταπολέμησης της απάτης και με αρχές οι οποίες, σε χώρες οι οποίες είναι σε προενταξιακή διαδικασία. Υπήρξαν διαδικασίες ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες σίγουρα είχαν πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο και μας ε, προσέφεραν πρέπει να πω και εξαιρετικά αποτελέσματα από πλευράς ε, ε συνεργασίας. Πολύ γρήγορα γιατί μετά ε, ο ε, στρατηγός Τόσκι θα μπορέσει να σας μιλήσει γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε, ίσως θα πρέπει να το είχαμε πει και από την αρχή, και πόσο σημαντικά έχει δραστηριοποιηθεί η μονάδα αυτή σε εθνικό επίπεδο κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία της πρόληψης αλλά και της ανάκτησης ποσών. Ε, η έμφαση ε, στην πρόληψη δόθηκε σκεμμένα διότι ε, διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο τομέα να εργαστούμε με πολύ μεγάλη πεποίθηση για να προλάβουμε τον κίνδυνο παραβιάσεων διότι η ανάκτηση των ποσών είναι πολύ πιο δύσκολη στη συνέχεια και η τιμωρία στη συνέχεια είναι τελείως διαφορετική. Είναι πολύ δύσκολο να κτίσει κάποιος ποσά από παράνομες δραστηριότητες και σε πρακτικό επίπεδο, σε πρακτικό διοικητικό επίπεδο. Επομένως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, αλλά και πολύ μεγάλη έμφαση ε, στην ε, κατάρτιση. Κατάρτιση της δημόσιας διοίκησης, κατάρτιση και σε περιφερειακό επίπεδο, διότι κυρίως ε, στη δική μας την περίπτωση της Ιταλίας οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ανάκτηση των ποσών, ιδίως όταν πρόκειται για ε, ποσά τα οποία φορούν την πολιτική συνοχή ή γεωργικά ταμεία. Πρέπει λοιπόν να είναι κατάλληλα καταρτισμένες οι διάφορες δομές της δημόσιας διοίκησης στα διάφορα επίπεδα και πάρα πολύ μεγάλη ε, δέσμευση σε επίπεδο ψηφιοποίησης ε, της και μηχανοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, διότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει κάποιος ειχνηλασιμότητα και πολλές φορές ε, ε, σε διασυνοριακό επίπεδο πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος κάποιες παρανομίες. Πρέπει κάποιος να διαθέτει στοιχεία. Στοιχεία τα οποία θα μπορούν να συγκρίνουν από εκεί και πέρα οι εθνικές αρχές, να τα διαβουλευτούν και να ανταλλάζουν και τέτοια στοιχεία. Μία πολύ σύντομη αναφορά στα γενικά στοιχεία πριν ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. η δραστηριότητα αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται σε μια σειρά από προτεραιότητες οι οποίες προωθούνται με ιδιαίτερη πειθό από τις Ιταλικές αρχές. Εμείς ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της απάτης, αλλά επίσης πολλαπλασιάσαμε και τις προσπάθειές μας στις διαδικασίες επί παραβάση. Έχουμε μειώσει ε, κατά το ίμιση τις διαδικασίες επί κατά της Ιταλίας και έχουμε ε, αυξήσει και τις προσπάθειές μας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Προσπαθούμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή επικρίσεων για την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ανταγωνισμού. Το κάναμε καταρχάς διότι αυτό είναι το σωστό, να υπάρχει κατάλληλος συντονισμό των εθνικών δραστηριοτήτων και να συντάσσονται και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το κάναμε επίσης και γιατί είμαστε βέβαιοι ότι αν θέλουμε να ζητήσουμε κάποια πράγματα από την Ευρώπη σε επίπεδο πολιτικών θα πρέπει ε, πρωτίστως να παρουσιάσουμε και τα διαπιστευτήριά μας και να δείξουμε ότι υπάρχει συνέπεια σε αυτό που κάνουμε. Και το κάναμε και γιατί είμαστε πεπισμένοι και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης ε, ότι το δίκαιο, η ακαιρεότητα του δικαίου, το κράτος δικαίου είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη γενικότερη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εάν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την νομιμότητα σε όλες τις μορφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ένας οργανισμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα περιέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση. Επομένως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων μας που ε, κάνουμε εμείς στις διαδικασίες επιπαραβάσεις, το τομέα της καταπολέμησης της απάτης και άλλες πολιτικές τις οποίες προωθούμε ε, ταυτοχρόνως, όπως για παράδειγμα τις πρωτοβολίες υπέρ του κράτους δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι συνδέονται με το ίδιο νήμα ε, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πρόγραμμα ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μελών και δράζεται αυτό στο κράτος δικαίου και στην καταπολέμηση οποιασδήποτε παράνομης ε, και άτυπης χρήσης των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και των κονδυλίων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο νομιμότητα νομιμότητας και της ε, προάσπισης του δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους παρισταμένους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, ε, στρατηγό Τόσκι και τον στρατηγό Ατάρδη για τα όσα έχουν κάνει ε, την Σύμβουλο Γκώση η οποία είναι εδώ διότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα αυτό και θέλαμε να την παρουσιάσουμε και εδώ στην Επιτροπή σας και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να σα πω από την πλευρά τη Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού. Ε, χαίρομαι το γεγονό ότι η Ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει πραγματικά ασκήσει πολύ αξιόπιστα αυτή τι προσπάθειε τη καταπολέμηση τη απάτη και δεν μπορούμε να το πούμε για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, και τη συμπερίληψη του του τη θεμένη αξία, έχει κάνει περισσότερε προσπάθειε. Θεωρώ λοιπόν πω ε, πραγματικά ε, θα ήταν δυνατόν να είχαμε επιτύχει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα και μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα αποτελέσματα με την Ιταλία από ό,τι σε σχέση με άλλα κράτη ε, μέλη. Δίνω όμως τώρα το λόγο στον του κ. Ατάρη. Καλησπέρα σε όλου. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αρχές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Είμαι ο στρατηγό Φραντσέσκο Ατάρντι ε, διοικητής ε, της μονάδας της Guardia di Finanza στο τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής ε, του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές που μας τιμούν με την παρουσία τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να χαιρετήσω και τον ε, κύριο Υπουργό, τον κύριο Νικόλα Βέρολα, ο οποίος είναι υφυπουργό αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και επικεφαλής της ε, τεχνικής γραμματείας ε, σε θέματα ευρωπαϊκών θεμάτων και την κυρία Ντιάνα Αγκόστο από το γραφείο του Πρωθυπουργού. η μονάδα της οποίας έχω την τιμή να βρίσκομαι επικεφαλής βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ε, βάσει συγκεκριμένη νομοθεσία είναι η τεχνική γραμματεία τη Επιτροπής, ε, της Εθνική Επιτροπή Καταπολέμηση τη Απάτη. Η Επιτροπή αυτή συστήθηκε το Φεβρουάριο του, του 1992 και από εκεί και πέρα συμπεριλήφθη στο οργανόγραμμα του Γραφείου του Πρωθυπουργού το Δεκέμβριο του 2012 συμμετέχουν στην Επιτροπή εκπρόσωποι στο υψηλότερο επίπεδο από όλες τις αρμόδιες αρχές στα θέματα αυτά και από πλευράς ε, διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και από πλευράς ελέγχων. Υπάρχουν ε, ε, δραστηριότητες οι οποίες είναι συμβουλευτικές ε, και συγκεκριμένες για το συντονισμό όλων των εθνικών και περιφερειακών ορχών που ασχολούνται με θέματα καταπολέμησης απάτης και παρατυπιών που αφορούν τον φορολογικό τομέα, την κοινή γεωργική πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρόκειται λοιπόν για το ιδανικό μέσο για την ανάλυση των παράνομων δραστηριοτήτων και για να βρούμε και ποιε είναι οι κατάλληλε στρατηγικέ για να μπορέσουμε να προβλέψουμε, να αντιμετωπίσουμε και να ε, ε αναστείλουμε τα συγκεκριμένα φαινόμενα παρατυπία και απάτης. Επίσης, ε, προσφάτως, ε, λάβαμε και τον τίτλο τη Κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμηση τη Απάτη. Ε, βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού 883 του 2013, τον οποίο θα αναφέρω στη συνέχεια και θα σας πω για ποιον ακριβώς λόγο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας κανονισμός ο οποίος υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να διαθέτουν μια υπηρεσία συντονισμού κατά πολέμηση της απέτης για να μπορέσουν να διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και επιχειρησιακής φύσεως ε, με την Όλαφ. Επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω ότι αυτό το άρθρο 3 περιλαμβάνει μια πρόταση την οποία προώθησε η Ιταλία σε μια συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Καταπολέμησης Απάτης της Κοκολάφ το ΙΟ του 2008. Οι Ιταλοί πρόσωποι πρότειναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσταθούν σε όλα τα κράτη-μέλη ένας οργανισμός κεντρικού συντονισμού καταπολέμησης απάτη, όπως ε, ε, κάνει σε εθνικό επίπεδο η Ιταλία. Τι κάνουμε, πώς συνεργαζόμαστε. Οι δραστηριότητες ε, τίθενται σε δύο επίπεδα, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τη συμμετοχή στις εργασίες της Ομάδας Καταπολέμησης Απάτης, της ΓΑΦ, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συντονισμού Καταπολέμησης Απάτης, της ΚΟΚΟΛΑΦ. Ε, δηλαδή το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη μέσω των εκπροσώπων τους συζητούν τα βασικά θέματα καταπολέμησης απάτης και τις ε, στρατηγικές ε, δράσεις που θα προωθήσουν σε κοινό επίπεδο. Επίσης, ε, η μονάδα αυτή δραστηριοποιείται και παρέχει υποστήριξη για τις ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή πληροφοριών και ειδήσεων στον Όλαφ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αρμόδια για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωσης. Επίσης ασχολείται με δραστηριότητε εταιρική σχέσης με τις αρμόδιες αρχές καταπολέμησης απάτηση των άλλων ευρωπαϊκών χωρών κυρίως ανταλλαγή εμπειριών, ε, περιπτώσεων και καλών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, ακριβώ σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο, η μονάδα καταπολέμηση απάτηση εγγυάται την εκπόνηση και την έγκριση από πλευρά ΑΦΚΟ αρκετών ε, πολύ συγκεκριμένων εγγράφων που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο τη έκθεση. Για παράδειγμα, το ετήσιο ερωτηματολόγιο του πρώην άρθρου 325 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης συμμετέχει και σε αυτές τις τεχνικές συνεδριάσεις της ΚΟΚΟΛΑΦ και της ΓΑΦ για τις οποίες ε, ε, κατά περίπτωση γίνεται συντονισμός και διαμορφώνεται η λεγόμενη εθνική θέση στα θέματα αυτά. Σε εθνικό επίπεδο, η Μονάδα Καταπολέμησης Απάτησης παρακολουθεί τις ροές επικοινωνίας που αφορούν περιπτώσεις παρατυπίες ή απάτης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ε, διαχειρίζεται εξ ονόματος της Όλαφ ε, ε, μία βάση δεδομένων, ένα σύστημα το οποίο αποκαλείται IMS, Irregularities Management System, ε, το οποίο ε, τους φέρνει σε επαφή με όλες τις αρχές διαχείρισης και σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, ε, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή αυτής της βάσης δεδομένων. Να προσθέσω απλώς εδώ ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να γίνει πολύ πιο καλή εφαρμογή, ε, επεκτάθηκε και ένα δίκτυο ε, για να υπάρχει ένα σημείο αναφορά σε όλες τις ε, αρμόδιες αρχές και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο για να έχουμε διευκόλυνση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανταλλαγής πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών και να υπάρχει έγκαιρη παρακολούθηση των διαδικασιών και να υπάρχει και επίλυση και κάποιων προβλημάτων ή κάποιων επικρίσεων. Για να σας δώσω μια ιδέα Επιτρέψτε με να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την εθνική επικράτεια έχουμε πάνω από 300 χρήστες, από τους οποίους ε, μόνο για το 2017, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, η μονάδα μας ε, πρόσφερε υποστήριξη σε πάνω από χίλιες ε, υποθέσεις περιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος ή για τα αιτήματα συνδρομής από τις αρμόδιες ε, Μια άλλη πολύ σημαντική ε, πτυχή, την οποία δεν θα πρέπει να υποτιμούμε, είναι ε, όλα όσα γίνονται σε επίπεδο προστασίας με τις εθνικές αρχές και των περιφερειακών αρχών για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και καθάρισης των ε, περιπτώσεων παρατυπιών ή απάτης, ε, οι οποίες πρέπει ε, να αφορούν κατά βάση την ανάκτηση των ποσών. Πρέπει να σας πω ότι εάν δεν επιληθούν το πρόβλημα, η κάθε χώρα ε, κινδυνεύει να έχει διπλή επιβάρυνση, γιατί αν δεν επιληθεί ε, θα τα χρεωθεί αυτή. Μια τελευταία δραστηριότητα είναι η συνεχής δραστηριότητα κατάρτισης για τα θέματα καταπολέμησης της απάτης των διαφόρων αρχών ελέγχου και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, ε, αρχές διαχείρισης, ελέγχου κλπ. Ε, και με επισκέψεις επιτόπου στις διοικήσεις για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε και την κάθε διαφορετική ε, περίπτωση. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που σας ανέφερα αναφέρονται στην ε, έκθεση η οποία υποβάλλεται κάθε χρόνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Μία έκθεση η οποία επισημαίνει τη λεγόμενη Εθνική Στρατηγική Καταπολέμησης Απάτησης ε, και ε, στο ιστορικό περιλαμβάνεται και μία αναλυτική ανάλυση κινδύνου με βάση την επεξεργασία όλων των στοιχείων για τις διάφορες περιπτώσεις παρατυπίας ή απάτης και χαράσονται και οι συγκεκριμένες στρατηγικές ε, γραμμές δράσης, δηλαδή οι δράσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν και οι στόχοι που θα επιτευχθούν ε, στα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένω, ε, η έκθεση περιλαμβάνει στα στατιστικά στοιχεία πάρα πολλά διαγράμματα και πίνακε που αναλύουν και πελιετέ περιόδου ε, και που αφορούν την εξέλιξη του πλαισίου όσον αφορά τι παρατυπίε και την απάτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και γίνεται και μια διάκριση ανατομέα ενδιαφέροντο. Και τι προκύπτει από όλα αυτά και από τη διαφάνεια που μπορείτε να δείτε. Προκύπτει ότι ο, ο ο οποίο πλήττεται περισσότερο είναι ο τομέα των των διαθροτικών ταμείων και των ταμείων επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 70% περίπου, ε, κάτι το οποίο ε, επιβεβαιώνεται πλήρως και από τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Ιταλία, στα οποία η παραβίαση ε, των, όσων αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, δυστυχώς πρέπει να σας το πω εγώ, αγγίζει το 80%. Και επίσης υπάρχουν και ε, σιγά σιγά ε, ε, περιπτώσεις ε, της λεγόμενης ε, διασυνοριακής απάτης, δηλαδή από οικονομικούς φορείς οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα οποία βεβαίωσε και η Όλαφ πρόσφατα στις τελευταίες εκθέσεις, κυρίως το 2016, η οποία μας είπε ότι αυτό το πρόσφατο φαινόμενο της διασυνοριακής απάτης αφορά ε, την ανάγκη να γίνουν κατεπηγόντως τροποποίησεις και αλλαγές στο παρόν ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάντησης. Ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή αφενός, επιτρέψτε μου να πω ότι εξακολουθεί ε, να έχει ε, σημαντική διαφορά σε κάθε χώρα και από την άλλη χρειάζεται πραγματικά ε, μια αποφασιστική ενίσχυση δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των ε, ερευνητικών οργανισμών της κάθε χώρας. Ακριβώς λοιπόν λόγω αυτών των επικροήσεων που μόλις αναφέρθηκαν, η στρατηγική δράση καταπολέμησης απάτησης της δικής μας υπηρεσίας της ΑΦΚΟΣ ε, επικεντρώθηκε κυρίως ε, σε ανταλλαγή, ε, αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών με όλες τις υπόλοιπε χώρες μέλους και να προωθήσουμε επίσης και συγκεκριμένες κοινέ δράσεις μέσω της καθοδήγησης και της Όλαφ. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος και είμαστε και όλοι πεπισμένοι ότι αν θέλουμε να διαπιστώσουμε τις περιπτώσεις απάτης και κυρίως να αποφύγουμε εγκαίρως να μην υπάρχουν παρανομίες, πρέπει να υπάρχει ένα ερευνητικό όργανο για την περίπτωση, για παράδειγμα, που θα πρέπει να εμβαθύνει αν πραγματικά υπάρχει κάποιο τιμολόγιο σε κάποια περίπτωση, να μπορεί ε, να απευθυνθεί στον ε, συνάδελφο για να δει τι δραστηριότητες έχει ε, ο οικονομικός φορέας, αν όντως υπάρχει πραγματικά κάποια δράση η οποία πρέπει να τιμολογηθεί κλπ. Και όπως προηγουμένως είπε ο, ο Υφυπουργός, η ΑΦΚΟΣ αποφάσισε να υποστηρίξει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία λήψη αποφάσεων μέσω ε, του λεγόμενου Cooperation Project in the Anti-Fraud Sector του 2016, το οποίο περιλαμβάνεται στη δημοσίευση που μεταξύ άλλων σας έχουμε παρουσιάσει σήμερα. Περιληπτικά, όλοι οι εμπειρογνώμονε των 15 χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμά μα ε, κατά την ε, ε, κατάρτιση του προγράμματο συμφώνησαν στο γεγονό ότι πολλά από τα προβλήματα σε θέματα πρόληψη και αντιμετώπιση τη διασυνορική απάτη έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Το γεγονό ότι δεν υπάρχουν κανόνε που μπορούν να επιτρέψουν να υπάρχει συγκεκριμένη και αποτελεσματική διοικητική συνδρομή στον ε, συγκεκριμένο τομέα των ε, ταμείων και των ταμείων επενδύσεων. Ε, υπάρχει λύση. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε βρει μια λύση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει να προλάβουμε το φαινόμενο της ε, απάτης ε, στον προπολογισμό της Ένωσης ε, και αυτό είναι η βελτίωση και η διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και αυτό φυσικά μπορούν να βρουν ε, να γίνει μέσω των αντίστοιχων ε, συντονιστικών μονάδων, των αντίστοιχων αύκοτ στις κάθε χώρα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Πέρσι αυτά τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε μια τελική διάσκεψη που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και ήταν παρόν εκεί και ο πρόεδρος Ταγιάννη αλλά και ο κύριος ε, Τόσκι, ο γενικός ο διοικητής μας αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές οι οποίοι θέλησαν να ε, επιβεβαιώσουν και ευχαριστούμε γι' αυτό ε, το ενδιαφέρον τους και για τη σημερινή συνεδρίαση. Και πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη ε, περηφάνεια διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για τα σχέδια της Επιτροπής ε, ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, αλλά και της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στο σημείο 50 του τελευταίου ψηφίσματος που πέρασε στις 16 Μαΐου, το αποδεικνύει αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε στο σημείο 50 το κείμενο, το οποίο λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε τα συμπεράσματα κλπ. Και εκεί προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ως ε, σημείο κίνησης ε, την ενδιάμεση αναθεώρηση που έγινε για την εφαρμογή του κανονισμού του 883 που ανέφερα στην αρχή της παρέμβασή μου που αφορά τις έρευνες που γίνονται από την Όλαφ. Επιτρέψτε μου τώρα εδώ να εκφράσω την ελπίδα ότι η Επιτροπή σας θα μπορέσει το συντομότερο δυνατό να συνεχίσει ε, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη τις αυτές τις ελπίδες και να χρησιμοποιήσει και την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του κανονισμού 883 του 2013 μέσω πιο στενής συνεργασίας των κρατών μελών και εκμεταλλευόμενη το δίκτυο επαφών που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, τον λεγόμενο ΣΑΦΚΟΣ των Κεντρικών Υπηρεσιών Συντονισμού της Καταπολέμησης της Απάτης. Ε, ολοκληρώνω λέγοντας ότι ακριβώς προκειμένου να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις και τις γνώσεις μας μεταξύ των ε, διαφόρων υπηρεσιών, τον ΑΦΚΟΣ, η Επιτροπή μας ε, εκπονεί ένα νέο σχέδιο συνεργασίας, όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός Βερολάν, και θέλουμε να το αναφέρουμε Cooperation Project 2 για να γίνεται ανταλλαγή ε, εμπειριών που έχουμε από έρευνες και να τεθούν και οι βάσεις, ε, και αυτό είναι μια καινοτομία, για τις λεγόμενες κοινέ ε, επιχειρησιακές δράσεις. Δηλαδή, ταυτόχρονες επιχειρησιακές δράσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα φαινόμενα της διασυνοριακής απάτης. Αυτό θα γίνει και σε πλήρη συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στο συγκεκριμένο ετήσιο ψήφισμά του, στο σημείο 90, ε, προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση των κοινών επιχειρησιακών δράσεων. Σε εθνικό επίπεδο, τι κάνει τώρα η ΑΦΚΟΣ ενισχύει περαιτέρω τις δραστηριότητες της εφαρμόζοντας ε, την διαδικασία της πρόληψης ε, της απάτης μέσω της ε, ε, δραστηριότητας μιας συγκεκριμένη ομάδας εργασίας ε, που οδήγησε στη δημιουργία μιας πλατφόρμας πληροφορικής για την καταπολέμηση της απάτης. Στις προηγούμενες εβδομάδες καθορίστηκαν πρακτικές πτυχές για την υλοποίηση αυτής της βάσης δεδομένων μέσω της στήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και θα ξεκινήσουν οι εργασίες πολύ σύντομα. Θα συνεργαστούν επίσης οι δράσεις για το προγραμματισμό, για τις πιο συχνές περιπτώσεις παρατυπίας και απάτης και το συγκεκριμένο τρόπο εργασίας ε, τον Σεπτέμβριο, όπω είπε προηγουμένω ο υπουργό Βέρολα, ξεκίνησε η νέα δέσμη μέτρων κατά πολέμηση απάτη, την οποία θέλαμε να μοιραστούμε με το Τμήμα Πολιτικών συνοχή του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Δικαιοσύνη, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εθνική Αρχή Κατά πολέμηση τη διαφθορά. Αυτό προβλέπει και συνεργασία με διάφορε περιφερειακές αρχέ για να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα εμβαθύνουμε όσον αφορά την πρόληψη και τη μετώπιση των παρανομών φαινομένων και επίσης να υπάρχουν συγκεκριμένε υποδείξει για τις διάφορες περιπτώσεις των πιο κοινών μορφών απάτης, ε, κυρίως στον τομέα των δραστηριοτικών ταμείων και να δούμε και ποιοι είναι οι δείκτε κινδύνου που θα μπορούσαν να επιτρέψουν ε, στους ε, υπαλλήλου που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους να διαπιστώσουν πολύ γρήγορα εάν υπάρχει απόπειρα απάτης ή παρατυπίες ε, και κατασπατάληση των δημοσίων πόρων. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά την ανάκτηση των ποσών και δυστυχώς ε, υπάρχουν επικρίσεις όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται για τον διαδικασία των ελέγχων. Υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από την ε, Αρχή Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Ταμείων στο Υπουργείο ε, πολιτισμού και τουρισμού και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη δράση συντονισμού για ένα λεγόμενο πρωτόκολλο συνεννόησης για να διευκολύνουμε και να δώσουμε κίνητρα για επιχειρησιακή υποστήριξη και γνώσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση ε, στο συγκεκριμένο τομέα των πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Και κάτι ακόμα, ε, και με αυτό ολοκληρώνω, διαδικασίες εξειδίκευσης για τον ευρωπαϊκών προγραμματισμών για κατηγορίες επαγγελματιών που θα μπορούσαν να θεωρούν ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον τομέα των ευρωπαϊκών ε, επιδοτήσεων, για παράδειγμα για λογιστές ε, ή σε κάποιες περιπτώσεις εξειδικευμένους νομικούς. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό ε, τομέα κλειδί για να μειώσουμε ουσιαστικά το λεγόμενο ποσοστό σφάλματος στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και μέσω ε, και της κατάρτισης συγκεκριμένων επαγγελματιών που ε, έχουν συγκεκριμένη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι ε, υπάρχει κάτι το οποίο για το οποίο μάλλον είμαι βέβαιος. Ίσως με την εμπειρία που είχαμε στην ε, ε, προηγούμενα χρόνια και επειδή έχουμε και συγκεκριμένη τεχνογνωσία θα μπορέσουμε στο εγγύς μέλλον να είμαστε ε, συγκεκριμένο εταίρος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων των αρχών καταπολέμησης απάτης των άλλων χωρών της Ένωσης με μόνο μία συγκεκριμένη προοπτική να έχουμε πραγματική προστασία των κοινών οικονομικών πόρων. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω λεπτομέρειες ε, μπορούμε να σας προσφέρουμε και έγγραφα και στοιχεία για τα θέματα τα οποία ανέφερα ακροθυγό σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ε, συνοπτική παρουσίαση. Ε, αλλά θα ήθελα να θέσω και ένα διευκρινιστικό ερώτημα. Ε, εδώ αυτά τα νούμερα που βλέπουμε είναι ποια είναι η πηγή τους, ευρωπαϊκή ή ιταλική. Είναι τα ευρωπαϊκά στοιχεία εντάξει, ότι σας κατάλαβα σωστά. Κύριε Σταδιέδε, έχετε εσεί τώρα το λόγο, παρακαλώ. Τόση. Κομισιόνε Κόντα del Parlamento Europeo. Σε του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχές ε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Καταρχάς, θα ήθελα να σα ε, ε, χαιρετήσω εγώ προσωπικά από πλευρά Guardia di Finanza και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση. Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται σε μια περίπλοκη και πολύ συγκεκριμένη διαδικασία προγραμματισμού και θεωρώ ότι είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία για τις στρατηγικές οι οποίες στόχο έχουν να εγγυηθούν μεγαλύτερη ασφάλεια σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσίευση η Cooperation Project in the Anti-Fraud Sector αποτελεί ουσιαστικά το άθροισμα των αποτελεσμάτων μια εις βάθος ανάλυσης η οποία είχε στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει την έγκριση ενός κανονισμού αμοιβαία διοικητικής συνδρομής η οποία θα γίνεται σε άμεσο επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Η πρωτοβουλία αυτή η οποία έγινε από την Επιτροπή Καταπολέμησης Απάτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δραστηριοποιείται στο γραφείο του Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Η Guardia di Finanza ε, έδωσε συγκεκριμένου πόρους ε, διότι είναι απόλυτα πεπισμένη ότι αν υπάρχει κανονισμό στον τομέα αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και εξοικονόμηση πόρων για να υπάρχει και διερευνητική δράση και θα έχουμε και περιγαλύτερη προσέγγιση και κοινά στοιχεία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα νομικό μέσο ε, συνεργασίας ε, σε διοικητικό επίπεδο και αυτό υποστηρίξαμε και στην διάρκεια του Ιταλικού Εξαμήνου της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ομάδα Καταπολέμησης Απάτης και την Προεδρία της ομάδας αυτής είχε εκπρόσωπο της Guardia του Finanza. Επίσης, η υποστήριξη στο έργο αυτό ε, συγκεκριμενοποιήθηκε και με τη συμμετοχή εκπροσώπων ε, της ε, διοίκηση και τη μονάδα τη Guardia di Finanza για την καταπολέμηση τη απάτη ε, κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ε, στι συναντήσει και στι ομάδε εργασία που οργανώθηκαν στα διάφορα στάδια τη πρωτοβουλία, ε, στη διάρκεια των οποίων μπορέσαμε να αναφέρουμε τι εμπειρίε μα, αλλά και να ανταλλάξουμε κοινέ τεχνικέ έρευνα. Επιπλέον, οι αρμοδιότητες της ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστυνομίας, τι οποίες χωρεί η Ιταλική νομοθεσία στην Guardia di Finanza, ε, σημαίνουν ότι η προστασία του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στόχος απόλυτης προτεραιότητας ε, της αποστολής του και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης δέσμευσης του τομέα των ε, δημοσίων δαπανών. Πρόκειται για μία δέσμευση η οποία ε, εδράζεται ε, σε πολύ παλιά χρόνια, διότι από το 1999 το Εθνικό Κοινοβούλιο ευθυγραμμίστηκε στις κοινοτικέ νομοθεσίε και ε, ανέθεσε στην Guardia τη Finanza το καθήκον να προλαμβάνει και να ε, ανακτά τις, τα ποσά από παράνομε δραστηριότητε των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια ενό ε, ευρύτερου πλαισίου επαγρύπνησης που σήμερα βρίσκεται στην Επιτροπή Καταπολέμησης Απάτησης το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που επιτρέπουν στην Guardia di Finanza να παρέμβει στον τομέα αυτό ε, διευρύνθηκε και τελειοποιήθηκε σταδιακά. Σήμερα όλα τα τμήματά μας έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν πέραν ε, του έργου τους ως ε, ε, δικαστική αστυνομία αλλά και σε διοικητικό επίπεδο και παρεμβαίνουν κατά της κοινοτικής απάτης ε, βάσει των ε, εξουσιών που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και από την νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανόμων εσόδων και αυτό φυσικά σημαίνει ότι η Ιταλία ε, ε, δίνει μεγάλη σημασία στην αρχή της προσωμίασης που αναφέρεται στο άρθρο 325 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη εγκρίνουν για να καταπολεμήσουν την απάτη που αφορά τα ε, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ίδια μέτρα τα οποία εγκρίνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των εθνικών οικονομικών συμφερόντων. Πρόκειται για ε, μεγάλη περηφάνεια για μας ε, το γεγονός ότι ο Εθνικός Νομοθέτης ε, θεώρησε ότι το αρμόδιο όργανο για την επιχειρησιακή δράση είναι η Guardia di Finanza. Πρόκειται για έναν, μια αρχή η οποία υπάρχει εδώ και 240 χρόνια. Η Guardia di Finanza για την καταπολέμηση της κοινοτικής απάτης ε, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο που αφενός έχει τον ε, διοικητή ο οποίος έχει την αποστολή να καθορίσει τις στρατηγικές ε, κατευθυντήριες γραμμές και να διευθύνει και να λαμβάνει υπόψη της τις θεσμικές σχέσεις αλλά και τις διεθνείς σχέσεις. Επιπλέον, η ειδική μονάδα για τις δημόσιες δαπάνες και την αντιμετώπιση της κοινοτικής απάτης, η οποία κατά προτεραιότητα ε, κάνει ανάλυση κινδύνου μέσω της διασταύρωσης των εσωτερικών βάσεων δεδομένων και των βάσεων δεδομένων εκτός Guardia di Finanza, τη μελέτη των συστημάτων απάτης, την εκπόδευση επιχειρησιακών μεθοδολογιών και την τεχνική και ε, πληροφορική υποστήριξη όλων όσων δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και η συμβολή του της λεγόμενης ειδική μονάδας για την ανάκτηση σε εθνικό επίπεδο των ε, καλύτερων εμπειριών που διαπιστώνονται επί τόπου μέσω των ε, λεγόμενων εργασιών βάση ε, έργου που αναπτύσσονται με την ε, στοχευμένη επιλοξή συγκεκριμένων επιχειρήσεων που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένα έργα έρευνας με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα. Πρόσφατα η μονάδα μας έχει και κάποιες συγκεκριμένε επιχειρησιακές δράσεις μέσω της σύστασης μιας ομάδας έρευνας ad hoc η οποία ε, έχει και τη δυνατότητα να κάνει απευθείας ε, έρευνες. Σε κεντρικό επίπεδο δραστηριοποιείται επίσης και η μονάδα της Guardia di Finanza για την ε, καταστολή της απάτης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιείται στο τμήμα στο Υπουργείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής που είναι ε, αρμοδιότητα του Υπουργού ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής και σε αυτό αναφέρθηκε ο στρατηγός Φρανσέσκο Ατάρντι. Σε επίπεδο περιφέρειας αυτή τη στιγμή σε όλες τις ε, διοικήσεις της περιφέρειας στα μονάδες της Guardia di Finanza υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα ή ομάδες για την προστασία της δημόσιας δαπάνης οι οποίες συνεχώς και μονίμως ασχολούνται με όλες τις υπηρεσίες αντιμετώπισης της κοινοτικής απάτης. Η ε, διαδικασία αυτή της περιφερειακής ε, μονάδας συμπληρώνεται και από και πολλές ε, διαφυγικές μονάδες, ομάδες, επιχειρήσεις, ε, τάγματα τα οποία ε, αποτελούν ε, τα διάφορες μονάδες της Guardia de Finanza. Οι δραστηριότητες μας κυρίως θέλουν να οδηγούν σε διαπίστωση ή παρατυπίας και που αφορά την γεωργική πολιτική αλλά και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο έλεγχος για την νομιμότητα των κοινοτικών ενισχύσεων καθορίζεται σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι να γίνεται εκ των ε, προτέρων έλεγχος, ο οποίος προηγείται της καταβολής της ενίσχυσης και στόχο έχουν να αξιολογήσουν κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση ε, στις αιτήσει που υποβάλλονται ε, με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την νομοθεσία για να δοθεί χρηματοδότηση. Το δεύτερο περιλαμβάνει τους εκ των υστέρων ελέγχους, οι οποίοι γίνονται μετά την εκταμίαση των κονδυλίων και, έχουν, και την ε, παράδοσή τους ε, στους δικαιούχους και αφορούν ε, την εκαθάριση των συγκεκριμένων παροχών και επιλέγονται βάσει συγκεκριμένης ανάλυσης κινδύνου όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και σας ανέφερα και προηγουμένως. Η τρίτη περίπτωση, στην οποία κυρίως αποτελεί αρμοδιότητα της Guardia da αφορά πιο συγκεκριμένε, πιο στοχευμένες δράσεις οι οποίες λέγονται έλεγχοι κατά πολέμηση απάτης οι οποίοι γίνονται βάσει υποψίας απάτης ε, που έχει διαπιστώσει είτε η αστυνομία είτε η δικαστική αστυνομία. Αυτή η κατηγορία των ελέγχων περιλαμβάνει ε, με συντονισμένο και συμπληρωματικό τρόπο και τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις που γίνονται βάσει των δύο προηγούμενων διαδικασιών. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, νομοθετικές διαδικασίες, οι οποίες ε, την τελευταία πενταετία ασχολήθηκαν με την ειδική μονάδα για τις δημόσιες διαπάνες και την αντιμετώπιση της κοινοτικής απάτης και έχουν διευρύνουν ε, τις αρμοδιότητες που μπορούμε να έχουμε στο τμήμα της δημόσιας δαπάνης και περιλαμβάνονται φυσικά και τα όσα αφορούν τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο πρόσφατη καινοτομία, η οποία εισήχθη από το ε, Προεδρικό Διάταγμα 83-2012, το λεγόμενο Διάταγμα Ανάπτυξης, ε, περιλαμβάνει την επέκταση των ε, εξουσιών ε, ε, κατά πολέμηση νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων όσον αφορά όλες τις δημόσιες δαπάνες. Στην Ιταλία έχουμε συμπεριλάβει τη κοινωτική δαπάνη στην ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που είναι ο κινητήριος μοχλός όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Το προσωπικό αυτή τη ειδική μονάδα που ασχολείται με τον τομέα τη δημόσια δαπάνη, αυτή τη στιγμή έχει και την αρμοδιότητα να ασκήσει τι εξουσίε που προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία από το ε, Προεδρικό Διάταγμα Διάταγμα 148-1988 που προβλέπει τη δυνατότητα να γίνονται έρευνες σε επιχειρήσεις και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, ή και σε άλλους ε, για τους οποίους ε, συντρέχει λόγος να θεωρείται ότι υπάρχει σχετική τεκμηρίαση πέραν της ιδιωτικής τους κατοικίας και να μπορούμε να ζητήσουμε να μας επιδείξουν λογιστικά βιβλία, έγγραφα, λιλογραφία και να λαμβάνουμε αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα οποιοδήποτε εγγράφου από αυτά που σας ανέφερα οι ίδιοι εξωματικοί μπορούν, ε, εάν θεωρήσουν ε, ότι συντρέχει λόγος, να διαβουλευτούν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στα φορολογικά στοιχεία που αφορούν και το αρχείο των σχέσεων με τους οικονομικούς φορείς. Πρόκειται λοιπόν για εξουσίες πάρα πολύ εκτεταμένες. Ε, βάσει της νομοθεσίες ε, και των ε, ε, επιχειρησιακών οδηγών, οδηγιών της Guardia di Finanza, οι εξουσίες οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή μπορούν να εκχωρηθούν στις αντίστοιχες μονάδες που έχουμε επιτόπου, είτε σε εδαφικό, είτε και σε λεγόμενες μονάδες της Guardia di Finanza. Ε, τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, κατά την άποψή μου, αποτελούν πολύ συγκεκριμένη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο προσπαθούμε εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτές τις πολύ σημαντικές ευθύνες. Χωρίς να ήθελα να επεκταθώ και να σας δώσω στοιχεία, θα ήθελα να περιοριστώ να σας υπενθυμίσω ότι από τον Ιανουάριο του 2015 και τους πρώτους 10 ε, μήνες του 2017 μετά από περίπου 7.000 παρεμβάσεις στον τομέα των ε, κονδυλίων του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώθηκαν απάτες και παρατυπίες για συγκεκριμένα αιτήματα και ε, ε, παρατυπίες στην ε, ε, στα κοινοτικά κονδύλια άνω των 900 εκατομμύριων ευρώ και πάνω από 500 εκατομμύρια αφορούν τα δραστηριοτικά ταμεία και τις άμεσες ενισχύσεις και 400 εκατομμύρια ε, τους πόρους της κοινή γεωργικής πολιτικής και της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Στο αντίστοιχο διάστημα, επαναλαμβάνω, Ιανουάριος 2015 και οι πρώτοι 10 του 2017, υπήρχαν καταγγελίες ε, στη δικαστική αρχή ε, άνω των 3.000 ατόμων. 30.000, 3.000 άτομα για απάτη, ε, κακοδιαχείριση και ε, λαθασμένη εκταμίαση κοινοτικών κονδυλίων και είχαμε δέσμευση εσόδων από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες άνω των 60 εκατομμύριων ευρώ. Φυσικά σε αυτό το πλαίσιο ε, δραστηριότητας η Guardia di Finanza και ως δικαστική αστυνομία αλλά και ως οικονομική χρηματοπιστωτική αστυνομία έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και όσον αφορά τη συνδρομή που η οποία παρέχεται για τις έρευνες που κάνει η Όλαφ για την προστασία της ε, δημόσιας ε, δαπάνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Όλαφ η ε, Guardia de Finanza έχει παραδοσιακά έντονη πολυετή και αποτελεσματική δραστηριότητα συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις συνεργασίας με την Όλαφ ευκρινίστηκαν ακόμα καλύτερα από το πρωτόκολλο συνεννόησης το οποίο μονογράφηκε το 2012 ε, το προηγούμενο, υπενθυμίζω και στον εαυτό μου υπογράφηκε το 1996, που καθορίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα ανταλλαγή πληροφοριών και επιχειρησιακών στοιχείων που θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τι συγκεκριμένε απαιτήσει και τις δικαστικές προτεραιότητες ε, να υπάρχουν τρόποι συνεργασίας, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επίσης να προλαμβάνουμε και αυτά τα οποία είχαμε ε, στη συνέχεια ε, στις διατάξεις του κανονισμού 883 του 2013 σε θέματα συνεργασίας μεταξύ Όλαφ και κρατών μελών. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ Όλαφ και των τμήματων του Σκουάρτια τη Finanza σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζεται και από το δεύτερο τμήμα της Γενικής Διοίκησης ε, μονάδα η οποία είναι αρμόδια για τις στρατηγικές ε, διεθνούς συνεργασίας ε, της Guardia di Finanza. Ο, έχουμε εδώ παρόν και το Γενικό Διοικητή, το Ρικάρντο Ραπανότη. Ε, ακριβώς λοιπόν αυτή η συνεργασία με το τμήμα αυτό ε, μας βοήθησε να εγγυηθούμε με πολύ σημαντική αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια πολλές επιχειρησιακές δράσεις, ε, συνεδριάσεις συντονισμού και στην Ιταλία και στο εξωτερικό για την ε, εκπόνηση στοχευμένων και πολύ συγκεκριμένων επιχειρησιακών παρεμβάσεων ε, με στη αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων ουσιαστικών αποτελεσμάτων αντιμετώπισης της απάτης όπως καταδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτό καταδεικνύει ότι η προτεραιότητα του δεύτερης μονάδας ε, της Guardia di Finanza έχει ως αρμοδιότητα να διασφαλίσει πιο αποτελεσματική και διαρθρωμένη ανταλλαγή μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Μια στρατηγική γραμμή ώστε η Όλεφ να έχει τις καλύτερες δυνατότητες να εκπονήσει την εντολή της ε, και Ελπίζουμε ότι ε, τα όσα προέκυψαν μετά από την έναρξη ισχύω του κανονισμού 883 του 2013 δεν επιτρέπεται βάσει του κανονισμού αυτού να ασκήσει αυτόνομα η όλα δραστηριότητες έρευνας στον τομέα αυτό και αυτό γίνεται λοιπόν από τις αρμόδιες αρχές. Ε, ακριβώς λοιπόν ε, λόγω των συνεργειών που καθορίστηκαν μεταξύ της Guardia de Financia και της Olaf επιβεβαιώνεται και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά καταρτίζονται ετησίως από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης, την Olaf και πολύ συχνά οι ερευνητικέ μεθοδολογίε τη Guardia di Financia και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει αναφέρονται στα έγγραφα ακριβώ λόγω αυτή τη σχέση. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ ε, συγκεκριμένα και στη συνεργασία μεταξύ Όλαφ και Guardia τη Φινάνσα στα θέματα προστασίας των εσόδων της Ένωσης, κυρίως στην καταπολέμηση ε, στο λαθρεμπόριο ε, τσιγάρων. Υπάρχουν πολλές διασυνοριακές έρευνες χάρη στην ουσιαστική συμμετοχή του Guardia di Finanza και είχαμε δέσμευση σημαντικών ποσοτήτων τσιγάρων στους λιμάνες και στα αεροδρόμια της Ιταλίας και επίσης καταφέραμε να ε, εξαρθρώσουμε οργανωμένα ε, ε, οργανωμένες κλιματικές μονάδες που ασχολούνται με αυτό το παράνομο εμπόριο. Τα στατιστικά στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένω, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη τη ιταλική δικαιοσύνη ε, στι δραστηριότητε τη Guarda di Finanza για να μπορέσει να εμβαθύνει για τα εναλλακτικά σενάρια για τι υποθέσει απάτη και κακοδιαχείριση των ε, κοινοτικών πόρων με προοπτική να έχουμε πραγματική ανάπτυξη, ανα, των ε, ποσών που έχουν ε, συσσωρευτεί. Εμπιστοσύνη η οποία προκύπτεται από, και από τη δική μας δυνατότητα να συνδυάσουμε τις τεχνικές ε, έρευνας που κάνει η Guardia di Finanza και να εμβαθύνει επίσης και σε θέματα τεκμηρίωσης ε, λογιστικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων ακριβώς λόγω των ερευνών που κάνουμε. Ε, βάσει λοιπόν αυτών των πολύ σημαντικών επιχειρησιακών εμπειριών, η Guardia di Finanza είναι απόλυτα πεπισμένη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα μέσο το οποίο θα ρυθμίζει την διοικητική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των διαφορετικών ταμείων. Ε, εξάλλου πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε ένα κενό το οποίο είναι και επικίνδυνο δεδομένου ότι ε, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι πόροι οι οποίοι προκύπτουν από αυτά τα συγκεκριμένα οικονομικά μέσα και υπάρχουν και κίνδυνοι ε, κακής ε, ε, χρήσης κυρίως από την, το οργανωμένο έγκλημα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο και διασυνοριακό σύστημα, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε και αποτελεσματικά μέσα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν στα όσα μπορούμε να έχουμε μέσω δικαστικής οδού, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο κατόφλι παρέμβασης ε, βάσει συγκεκριμένων ε, ενδείξεων που πρέπει ακόμα να ε, καθορίσουμε σε ποινικό επίπεδο. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή της συνεργασίας που προσφέρεται ε, από την Guardia di Finanza, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ και να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Guardia di Finanza βάσει και τις αποστολές ε, τις οποίες έχει αναθέσει ο Ιταλός νομοθέτης θα συνεχίσει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκειμένου να εγγυηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα την προστασία της νομικότητας των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων που είναι πολύ σημαντικός παράγον για την εγγύηση της ανάπτυξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στρατηγέ για αυτή την παρουσίαση. Ε, ποιο είναι το νήμα, αν θέλετε, ένα κοινό νήμα που διατρέχει και τις τρεις ε, παρουσιάσεις. Είναι η ελλειπής υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία. Έχουμε δημιουργήσει βέβαια κάποιες υπηρεσίες, για παράδειγμα την Όλαφ, έχουμε την Eurojust, και στο μέλλον θα έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία βέβαια θα χρειάζεται και πάρα πολύ σοβαρές υπόνες για να μπορεί να αναλάβει δράση αλλά από εκεί και μετά ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ε, να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα ως προς το ποια ακριβώς υποστήριξη θα μπορούσατε να λάβετε από τα Διευθυντικά ταμεία και σε τι είδους ε, δραστηριότητες θέλετε υποστήριξη, για παράδειγμα, ε, για την καταπολέμηση εγκληματικών οργανώσεων, ε, σε ό,τι αφορά παρατυπίες στο δημόσιο τομέα. Γιατί βέβαια η τέτοιου είδους υποστήριξη μπορεί να δοθεί, αλλά περιλαμβάνει και σημαντικές καθυστερήσεις. Κάτι ακόμα τώρα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Αδεπάτη στην Όλαφ. Ε, δηλαδή τα νούμερα που μας αναφέρετε εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακά. 3.000 άτομα μας είπατε σε, και 7.000 ε, παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα, τις ε, δαπάνες ε, κοντιλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 3.000 άτομα να εμπλέκονται σε αυτές τις 7.000 υποθέσεις. Άρα λοιπόν, σε όλες αυτές τις υποθέσεις ποιον ακριβώς ρόλο παίζει ο Όλαφ γιατί αυτή η συστηματικό, ο συστηματικός έλεγχος ε, που λαμβάνει χώρα ε, των δημοσίων ε, δαπανών και ο οποίος πραγματικά είναι ασύγκριτος. Δεν ξέρω ότι να υπάρχει κάποιο άλλο κράτος μέλος στον οποίο να προβαίνει σε ένα τέτοιο έλεγχο. Πώς ακριβώς λαμβάνει χώρα. Δηλαδή, πώς αξιοποιείται για παράδειγμα τις εκθέσεις της Όλαφ για να προβαίνεται σε αυτούς τους ελέγχους και στη συνέχεια να προβαίνεται ενδεχομένω και σε ε, διώξεις των εμπλεκομένων. Γιατί βέβαια έχει αναφερθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να καταστούν πιο σαφεί αυτές οι εκθέσεις τη Όλαφ έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ο κ. είπε ότι ε, θα πρέπει να αναλάβει και ηγετικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο αναλυτικότερα αυτή την, ε, αυτή την ηγετική θέση που θέλετε να αναλάβει, γιατί, αναλάβει, γιατί βέβαια στο ε, εγγύς ε, μέλλον θα κληθούμε να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό της Όλαφ. Οπότε Εκείνο που σας ρωτώ είναι, παρότι θα είναι βέβαια μια δύσκολη ε, διαδικασία αυτή η αναθεώρηση, ε, ποια λοιπόν στοιχεία θεωρείτε πως είναι απαραίτητα για να μπορέσει να αναλάβει ένα τέτοιο ηγετικό ρόλο η όλα. Για παράδειγμα δεν αναφερθείτε καθόλου στο ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος και στη μαφία. Ίσως θα μπορούσατε να κάνετε και μια ανοίξη ε, σε σχέση με αυτό το είδο εγκλήματο. Γιατί βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τα όσα κάνουμε, γιατί βέβαια έχουμε αποτύχει των εισαγωγικών στο παρελθόν. Οπότε έχετε το λόγο, δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει πρώτος το λόγο. και Σας Ναι, σας ευχαριστώ. Για την Όλαφ, όπως σας έλεγα προηγουμένως, Εμείς ε, είμαστε πολύ δραστήρια σε θέματα βοήθειας, συνδρομής, ε, στήριξης με τα διάφορα άλλα θεσμικά όργανα, κυρίως με την Όλαφ. Και κυρίως, ε, όπως ανέφερα, βάσει και του άρθρου 3, σημείο 4. Για την Όλαφ να σας αναφέρω τις τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν το 2017 κατόπιν προτροπής της Όλαφ. Ε, λάβαμε υπόψη μας μία σειρά από αιτήματα, πέντε αιτήματα φέτος από την Όλαφ, για την ε, διεξαγωγή στην Ιταλία των λεγόμενων επιτόπιων ελέγχων. Εμείς ε, ε, αυτές τις ε, αναθέταμε στη δεύτερη μονάδα, όπως ανέφερε ο κύριος Τόσκι, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο σκηνοθέτης όλης αυτής της διαδικασίας, αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα στα όλα αυτά όσα συμβαίνουν στην Κορία και από εκεί και πέρα όλα αυτά ανατίθεται στα τοπικά, στις τοπικές μονάδες που ασχολούνται με το θέμα. Ε, αυτό σημαίνει ότι η Όλαφ καταρχάς ε, είναι ευγνώμων γιατί γίνονται οι έλεγχοι αυτοί ορισμένες φορές και από κοινού με εκπροσώπους της Όλαφ που έρχονται στην Ιταλία αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, δράσαμε τελώς αυτόνομα. Τώρα, τι άλλο προσφέραμε εμείς όσον αφορά τη συνεργασία με την Όλαφ. Συμμετείχαμε στην εκπόνηση μιας σειρά εγγράφων για παράδειγμα στα πλαίσια της ομάδας εργασίας των ε, Practical Steps ε, Toward Drafting and Anti-Fraud Strategy κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική καταπολέμηση της απάτησης και ούτω καθεξής, ε, αντιμετώπιση στις ε, δημόσιες συμβάσεις της απάτης. Υπάρχουν δηλαδή μία σειρά από πληροφορίες οι οποίες φτάνουν από την Όλαφ και εμείς ε, τις εφαρμόζουμε στη χώρα μας, ε, δίνουμε φυσικά και τα σχετικά στοιχεία. Μέχρι τώρα ήταν πολύ σημαντική και η ικανοποίηση της όλα για τα σημεία αυτά. Και επίσης, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και την αντίκτυπο που έχουμε και ποιος είναι ο πιο συνήθις τρόπος ε, παράνομης οικειοποίησης ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς επιμένουμε στο σημείο αυτό και με την Όλαφ για να ξεκινήσει να δημιουργείται μια κοινή δράση αντιμετώπισης. Ποιες είναι οι πιο συχνές ε, περιπτώσεις. Ε, η χρήση τιμολογίων που στην πραγματικότητα αφορούν ε, ποσά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ε, πολλές φορές υπάρχουν ε, ψευδή στοιχεία για ε, συγκεκριμένα ε, στοιχεία ενεργητικού τα οποία υποτίθεται ότι διατίθενται για να μπορέσουν να ληφθεί χρηματοδότηση, την οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Ε, πλαστές αυξήσεις του επιχειρησιακού κεφαλαίου, τα οποία, οι οποίες γίνονται ad hoc για να μπορέσει να λάβει κανείς τη χρηματοδότηση. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένε ε, δραστηριότητες ε, με χώρες οι οποίες έχουν ε, χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς, προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ορισμένες φορές προσπαθούν να παρακολύσουν τις διαδικασίες για να μην μπορέσει κάποιος να δει τι συνέβη μέσα σε μια επιχείρηση. Ε, δεν γίνονται σεβαστές υποχρεώσεις για την ε, ε, εκταμίευση της χρηματοδότησης. Υπάρχουν μία σειρά λοιπόν από διάφορες περιπτώσεις τις οποίες παρακολουθούμε συνεχώς και κάθε φορά το συζητάμε και με την Όλαφ και τα επισημαίνουμε διότι πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτά είναι τα ουσιαστικά σημεία τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να υπάρχει μια δομή και σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δεν μπορεί ο καθένας να δρά ε, μόνος του. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις ε, τι οποίε μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε χώρα, αλλά θα πρέπει να δούμε και από κοινού, διότι έτσι θα είμαστε πιο ισχυροί. Προηγουμένω αναφέρθηκα και εδώ έρχομαι και να απαντήσω στην ερώτησή σα. Αναφέρθηκα σε κάποιες δράσεις οι οποίε δεν είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ των κρατών μελών για τα όσα γίνονται για την καταπολέμηση της απάτη. Και το βλέπουμε όλοι. Υπάρχει ανομοιογένεια, άρα δεν υπάρχει ισοδύναμη δράση αυτή τη στιγμή μεταξύ των ε, κρατών μελών της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης. Αρκεί να σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των λεγόμενων δικαστικών συστάσεων που ε, ε, κάνει η Όλαφ ε, βάσει των δραστηριοτήτων της κάθε χώρας. Νομίζω στην ετήσια έκταση του 2016 της Όλαφ, τα αποτελέσματα αυτών των συστάσεων που γίνονται προς τα κράτη-μέλη, ε, οι οποίες διακρίνονται σε ναι ή όχι, δεν ελήφθη καμία απόφαση από τη δικαστική αρχή ή ελήφθη απόφαση από τη δικαστική αρχή. Αν κάνουμε τα σύγκριση αναχώρα, περνάμε από το 0% στο 100% σε κάποιες περιπτώσεις. Φοβίζουν αυτές οι διαφορές. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει συντονισμό στις δικαστικές αποφάσεις. Ε, προσφάτως, όπως γνωρίζετε, το αντιμετώπισε η Όλαφ και προσπάθησε να το εμβαθύνει και να το συζητήσει και να δει για ποιο λόγο οι διάφορε δικαστικές αρχές των διαφόρων χωρών δεν δίνουν συνέχεια στις συστάσεις που κάνουν οι ίδιες οι αρχές και προσπάθησαν να τα συμπληρώσουν όλα αυτά σε ένα έγγραφο το οποίο έδωσε μια σειρά από στοιχεία σε μια γνωμοδότηση της Όλαφ. Ε, πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία, τα διαβάσαμε όλοι, δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά αυτό το οποίο με εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις Υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ Όλαφ και εθνικών αρχών κρατών μελών ε, και κάποια πράγματα θεωρούνταν ησυχητικά από την Όλαφ. Ε, υπήρχε τέτοιος χαρακτηρισμός. Δίνονται ψευδείς, για παράδειγμα, πληροφορίες στις αρχές διαχείρισης και αυτό ε, δεν θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό ε, στοιχείο από κάποιες εθνικές αρχές. Δηλαδή ουσιαστικά δεν δίνεται ιδέουσα προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται και πλαστά έγγραφα για να λάβει κάποιος χρηματοδότηση. Ε, οι ερευνητές της Όλαφ, ε, για παράδειγμα, θεωρούν κάποια πράγματα παρατυπίας και δεν τα θεωρούν αντίστοιχα παρατυπίες τα εθνικά υπουργεία. Ε, για παράδειγμα, οι ερευνητές της Όλαφ θεωρούν ότι τα πλαστά τιμολόγια είναι απάτη. Ενώ από πολλές χώρες θεωρούνται τιμολόγια τα οποία δεν ε, πληρώθηκαν από τους ε, ε αρμόδιους οικονομικούς φορείς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι σοβαρές παρατυπίες και κάποιες χώρες τα θεωρούν απλώς σφάλματα, τα θα χαρακτηρίζουν ως σφάλματα. Είναι πολύ περίπλοκο το πλαίσιο που μας παρουσίασε η Όλαφ, είναι ένα σενάριο που περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία και νομίζω το είπε και ο Υπουργό Βέρολα προηγουμένως, αναφέρθηκε στο σημείο αυτό. Αυτό οδήγησε την Ιταλία να γίνει η χώρα η οποία ε, δίωξε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα φαινόμενα που αφορούν τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το 2009-2016 είχε από τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ε, εκδόθηκαν και είχε το λεγόμενο indictment rate του 63%, πολύ υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 44%. Θεωρούμε ότι οι επιδόσεις αυτές είναι ε, διότι λαμβάνουμε υπόψη την ουσία των συστάσεων προς την Όλαφ και αυτό αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη τιμές. Και θα ολοκληρώσω ε, με αυτό που είπε και ο διοικητής μου. Μία ιδιομορφία της Ιταλίας, πέραν αυτού της ε, δικαστικής δυνατότητας των επιδόσεων, είναι το γεγονός ότι στην Ιταλία υπάρχουν διοικήσεις οι οποίες είναι πολύ πιο αποτελεσματικές σε θέματα καταπολέμησης της απάτησης ε, διότι υπάρχει η Guardia di Finanza, αυτό το ειδικό τμήμα της αστυνομίας που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Η ειδική αστυνομία μάλλον, όχι ειδικό τμήμα της αστυνομίας. Προσπαθούμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα της Ένωσης μέσω μια πολύ συγκεκριμένη δομής, ε, εύρωστης και ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λαμβάνει πολύ συγκεκριμένε προτεραιότητε έρευνα και έχει πολύ συγκεκριμένε εξουσίε. Εγώ λοιπόν προσωπικά είμαι τη άποψη ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό και πολύ συγκεκριμένο τρόπο τα πιο συγκεκριμένα φαινόμενα απάτη, πρέπει να οργανωθούμε με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά κυρίω με αποδοτικό τρόπο. Στην Ιταλία είναι σχεδόν δεδομένο και αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν όμως ανάλογες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως σας είπα μέχρι τώρα δεν ακολουθούν την ίδια άγουσα άλλες χώρες μέλη. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει όλα. Πρόσφατα, βάσει ενός συγκεκριμένου ερωτηματολογίου που επιστάλησαν σε όλα τα ευρωπαϊκά αύκος, προσπάθησε να λάβει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις πρακτικές ε, μορφές διεξαγωγής ε, των ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης σε κάθε χώρα. Ολοκληρώνω λοιπόν με αυτό και να πάρει το λόγο ο κύριος Τόσκι τώρα. Ευχαριστώ το στρατηγό Ατάρντι διότι νομίζω ότι απάντησε με λαμπρό τρόπο στην πρώτη ερώτηση και θα ήθελα να ολοκληρώσω με τέσσερις παρατηρήσεις όσον αφορούν τη συνεργασία από πλευρά Guardian de Finanza για να βελτιώσουμε τη διαδικασία τη συνεργασία. Όσον αφορά τη δικαστική αρχή, εμεί εξαρτώμαστε από τι δικαστικέ αρχέ και για επιχειρησιακού λόγου, αλλά κυρίω εμεί ε, παρέχουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και σε όλε τι δικαστικέ αρχέ την πλήρη αμέριστη συνεργασία μα ε, για την ε, διαχείριση οποιασδήποτε δραστηριότητα και βοηθούμε και παρέχουμε στις δικαστικές αρχές Και υπάρχει συγκεκριμένη αναγνώριση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, για την ε, αποτελεσματική συνεργασία για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και δικαστές ε, και υπαλλήλου και εργαζομένους όμως ή αστυνομικούς της δικαστικής αστυνομίας πολλών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά για να μπορέσουν να γνωρίζουν και αυτοί και να κάνουν κτήμα τους την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εμείς σε θέματα ερευνών, κυρίως σε οικονομικό χρηματοπιστωτικό επίπεδο, προκειμένου να μπορέσουμε να ε, διαπιστώσουμε ε, όλες αυτές τις απάτες. Όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες τώρα της συνδρομής προς τα διοικητικά όργανα, πέραν των όσων είπε ο στρατηγός Ατάρτη, μέσω της δεύτερης μονάδας της Γενικής Διοίκησης, που έχω ενισχύσει σημαντικά εγώ προσωπικά και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο. Ξεκινούμε νέε διεθνεί δράσει, όχι μόνο με όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρούμε ότι είναι και αδέλφια μα ε, και βρισκόμαστε στην ίδια επικράτεια, αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Ε, ο υποφαινόμενος ε, ορίστηκε κατόπιν υπόδειξη του Υπουργού Οικονομικών ε, στην ΣΥΑΤ εκ μέρου των ε, ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχα και θα συμμετείχω και στη συνέχεια στην Αργεντινή και στην Παραγουάη σε πρόσφατες συνεδριάσει της ΣΥΑΤ για να μπορέσουμε να έχουμε και σε αυτό το υψηλότατο επίπεδο ε, μια παρουσίαση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έγιναν στην Ιταλία κυρίως από την Guardia di Finanza. Και θα ολοκληρώσω, μου επιτρέπετε, με την ίδια σκέψη και χαίρομαι που είναι εδώ και η κυρία Κινίτσι, διότι το ίδιο είπα και στην ακρόαση και τη συνάντηση που είχαμε με την Ειδική Επιτροπή ΤΕΡ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γιατί στην Ιταλία η Guardia di Finanza μπορεί να παρέμβει και παρεμβαίνει ίσως περισσότερο από άλλες χώρες. Διότι εμείς ιστορικά έχουμε έναν εχθρό ο οποίος είναι δυστυχώς ε, ιδιαίτερα παρόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη μαφία και με όλες τις συμμορφές, την Καμόρα, την Τράγκετα κλπ. Εδώ και χρόνια λοιπόν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, τη συγκεκριμένη μορφή ε, διεθνούς εγκληματικότητας, η οποία ασχολείται με τα πάντα, με κάθε μορφή εγκλήματος και κυρίως ε, τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων ε, και γενικότερα το λαθρεμπόριο για να ε, πλουτίσει φυσικά. Εμείς λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρησιακές δράσεις οι οποίες ε, μας δίδαξαν ε, από οι μαέστροι αυτών των ε, τεχνικών, να υπενθυμίσω ο δικαστής Κινίτσι, ο δικαστής Φαλκόνε, ο δικαστής Πορσελίνο, και εγώ θα ήθελα να προσθέσω και έναν εισαγγελέα, έναν από τους πρώτους εθνικούς εισαγγελείς καταπολέμησης της ε, Μαφία, τον πρώην Λουίτζι Βίνια. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαέστροι στην καταπολέμηση τη Μαφία και τη Τρομοκρατία και μα δίδαξαν ότι κανένα έγκλημα δεν θα πρέπει ε, να παραμελείται, καμία έρευνα δεν θα πρέπει να ε, γίνεται πλημελός για, ακόμα και αν πρόκειται για κάτι ελάχιστο, το οποίο τελικά μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει ε, σε παράνομα κέρδη. Ε, τώρα, πού για πού προερίζονται αυτά τα παράνομα κέρδη, ε, προορισμοί που δεν μπορείτε να τους φανταστείτε. Ορισμένες φορές και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς και η Guardia di Finanza, που είναι οικονομική και χρηματοπιστωτική αστυνομία, και πρέπει να ενισχύσει ε, τα οικονομικά ε, και χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, διότι πρόκειται για ένα σώμα προστασία του προπολογισμού κυρίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένω και του εθνικού και τοπικού προπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε και τόσο δραστήριοι και ε, άρτια καταρτισμένοι και επιβεβαιώνω ότι είμαστε και πλήρω διατεθειμένοι και στο μέλλον ε, ω Guardia de Finanza με όλε μα τι μονάδε να συνεργαστούμε όχι μόνο με την Όλαφ αλλά και με όλου του οργανισμού και τα τις αρχές που ασχολούνται με την καταπολέμηση της ευρωπαϊκής απάτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και τους ομιλητές ε, για όλο του το έργο και εγώ σπούδασα στη Ρώμη και πάντα ήμουν θαυμαστή της ε, Guardia de Finanza και του εξαιρετικού αυτού οργανισμού που με ιδιαίτερη περηφάνεια κλήρωνε το έργο του και εγώ είχα ένα φίλο που εργαζόταν εκεί και μου έλεγε ότι ήταν πραγματικά η ελίτ των Ιταλικών αστυνομικών δυνάμεων. Τα όσα μας παρουσιάσατε σήμερα καταδεικνύουν ακριβώς αυτό. Σαφώς και εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερως το έργο σας. Η Ιταλία αποτελεί υπόδειγμα ε, καταπολέμησης και της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως αυτό που βλέπουμε ακόμα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι ιδιαίτερη και ευρύτατη εφαρμογή ε, των απατών τύπου καρουζέλ ε, με εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται από ε, την Ανατολή προς τη Δύση. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε ε, πλασματική αποστολή αυτών των τιμολογίων και το καθεξής. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σωστή κατάρτιση. Από την εμπειρία μου βλέπω ότι οι δικαστές και εισαγγελίες συχνά δεν έχουν ιδέα από αυτά τα πράγματα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, έχετε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης για τους δικαστές από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για να αυξήσουμε ε, τα επίπεδα κατάρτισής τους ε, σε αυτά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί πολύ συχνά υπάρχει καταδίκη ε, πρωτόδικη και μετά κατά την έφεση η καταδίκη αυτή ανατρέπεται εξαιτίας ε, τυπικών ε, σφαλμάτων σε ό,τι αφορά την ε, παράνομη αυτή δραστηριότητα. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων. Πολλές φορές όταν έχουμε συζητήσει τέτοια ζητήματα με τους οικονομικούς φορείς στην Τσεχία, βλέπω ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι δεν καταρτίζονται όπως πρέπει. Οπότε ε, προτίθεστε να προσφέρετε τέτοιου κατάρτιση σε άλλους ε, συναδέλφους. Κυρία Κινίτση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ιταλούς ε, καλεσμένους μας. Εμείς συναντηθήκαμε και προηγουμένως σε μια ανεπίσημη συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής ΤΕΡ, της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία και τώρα είχα τη χαρά να τους παρακολουθήσω και εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω διότι παρουσίασαν ε, με σαφή ε, και ακριβή τρόπο την τεράστια δουλειά που γίνεται στην Ιταλία από την Guardia di Finanza σε γενικότερα θέμα αντιμετώπισης ε, της οικονομικής απάτης και σταθήκαμε και στον τομέα της απάτης για τα διαρθρωτικά ταμεία που είναι ίσως και ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο στρατηγός Τόσκι και ο στρατηγός Ατάρντι ε, απάντησαν στις ερωτήσεις ε, που ε, μου δημιουργήθηκαν, κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ της νομοθεσίας των διαφόρων χωρών και το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στη συνεργασία. Μου άρεσε η ιδέα μιας άμεσης διοικητικής συνεργασίας μέσω συντονισμού της Όλαφ, αλλά σε μία απόπειρα να γίνουν όλα ένα και πιο αποτελεσματικά ε, και πιο γρήγορα, να είναι πιο γρήγορε οι διαδικασίες και διάφορε επιχειρήσει. Έχω όμω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η συνεργασία, αναφέρθηκε και ο συνάδελφος προηγουμένω, κατά την άποψή μου βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και η αμοιβαία εμπιστοσύνη γεννιέται και από τη γνώση της δουλειά του καθενό και φυσικά και από την ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση. Δεν αρκεί μία κατάρτιση πολύ προσεκτική σε μία χώρα. Κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει ενιαία κοινή κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτό ε, σε συνδυασμό και με ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να δώσει μια περαιτέρω όθηση και κίνητρο για συνεργασία, αυτό το οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσον θεωρείτε ότι όταν αναφερόμαστε σε κατάρτιση θα πρέπει λίγο να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να αναφερθούμε σε μια κατάρτιση για όλες τις χώρες, ε, μια κατάρτιση ε, κοινή ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική συνεργασία. Και όσον αφορά το θέμα των ε, εγκληματικών οργανώσεων, ο κύριος Τόσκι ε, ε, απάντησε στην πραγματικότητα, αλλά όσον αφορά την Ιταλική εμπειρία, για αυτές τις μορφές εγκλημάτων μας είπατε εσείς ότι ορισμένες φορές τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες χρησιμεύουν για να χρηματοδοτήσουν πολύ πιο σημαντικές και πιο παράνομες διαδικασίες. Αυτό είναι ιδιαιτερότητα της Ιταλίας, το να χρησιμοποιούνται δηλαδή έσοδα από μία εγκληματική δραστηριότητα για να χρηματοδοτήσουν άλλες χειρότερες ή είναι ιδίων και άλλων χωρών. Και επίσης, εγώ πιστεύω και ε, πέραν της ε, ε, δράσης στην πρόληψη. Και νομίζω ότι ο στρατηγός Ατάρτ αναφέρθηκε στην, Ατάρτη αναφέρθηκε στην πρόληψη. Η ερώτηση είναι λοιπόν προς τον εαυτό μου, αλλά θα την απευθύνω σε εσά. Ίσως εμείς, κυρία Γκρέσλε, θα μπορούσαμε ως Κοινοβούλιο να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μνημόνιο πρόληψης, το οποίο θα μπορούσε να είναι κοινό, να υπάρχουν κοινά προγράμματα πρόληψης, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκές χώρες. Λίγο στις γραμμές του προγράμματος που μας παρουσίασε ο στρατηγός Ατάρτη και να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα πρόληψης και για την ιδέα αυτή που θα μπορούσαμε ίσως να προωθήσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το προτείνουμε σε όλες τις χώρες να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα πρόληψης στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Kollege Valli, bitte. Oh. Sì, un'altra Μία ερώτηση ακόμα, ο κύριος Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους στρατηγούς εδώ για την πολύ σκληρή δουλειά που κάνουν στη χώρα μας, αλλά και για ό,τι κάνουν ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προσπαθήσουν να προωθήσουν και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, γιατί και το κίνημα των πέντε αστέρων, που ορισμένες φορές ε, είναι ε, ευρωσκεπτικιστές ε, σε διάφορα θέματα. Όσον αφορούν την καταπολέμηση της απάτης, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ευρεία συνεργασία και διεθνής μάλιστα συνεργασία και χαίρομαι που υπάρχουν και διεθνείς μηχανισμοί για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Το Κοινοβούλιο πολλέ φορέ έχει εκφράσει την άποψή του υπέρ τη ανταλλαγή πληροφοριών για τα διαρθρωτικά ταμεία για τη σχέση των, ε, της προστασίας των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω τα κράτη-μέλη να τα λάβουν υπόψη τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εμπειρίες τις δικές μας. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές είναι πολύ προοδευτικό, αλλά στα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζονται όλα αυτά. Όσον αφορά τη διαφάνεια, η οποία κατά την άποψή μου είναι το θεμελιώδες ζήτημα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μορφή ε, της ε, ε, διασυνοριακής απάτης ε, στον τραπεζικό κόσμο θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η νομοθεσία σήμερα σας επιτρέπει να επαληθεύσετε και να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε μέσω διεθνών τραπεζικών ροών ή υπάρχουν κενά και εκεί και πρέπει να γίνει κάτι και στον τομέα αυτό. Διότι έχω την εντύπωση και στην όλη ευρύτερη συζήτηση για το ξέπλυμα χρήματο διεθνώ, ε, για του φορολογικού παραδείσου που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εδώ το Κοινοβούλιο, ότι οι μεγάλε τράπεζε, κυρίω οι μεγάλε επιχειρηματικέ τράπεζε, οι οποίε ε, από ό,τι διαπιστώνουμε και από τα διάφορα σκάνδαλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι ε, κάνουν ξέπλυμα ε, δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμες. Ε, μπορεί ο νομοθέτης εδώ να σας βοηθήσει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες επιδεικνύουν λιγότερη συνεργασία και αρνούνται να συνεργαστούν. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης συνεργάζονται ή όχι. Διότι πολύ συχνά για πάρα πολλά πράγματα ε, πολλές φορές ηθικολογούν αλλά δεν ξέρω κατά πόσον όσον αφορά την παραποίηση στους μεγάλους λιμένες της Ευρώπης δείχνουν οι ίδιοι πνεύμα συνεργασίας Κυρία Τζουφρίτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για την παρουσία τους εδώ και για την πληθώρα των πληροφοριών που μας έδωσαν. Και πρέπει να πω και για το τιτάνιο έργο το οποίο υλοποιούν, ε, το οποίο ας το πούμε και με κάποια εθνική περηφάνεια η χώρα μου πραγματικά ε, ηγείται ε, στον τομέα αυτό, στην αντιμετώπιση της απάτης ε, και ε, την ε, προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποια στοιχεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου. Το πρώτο αφορά τη μεγάλη προβολή του φαινομένου της απάτης, το οποίο σχετίζεται και πάρα πολύ στενά με την έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά και την απομάκρυνση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η οποία αυξάνεται συνεχώς. Πολύ συχνά οι ειδήσει που αφορούν ε, είτε αληθινές είτε ε, ψευδείς απάτες και θέματα που αφορούν τον τομέα της απάτης ε, χειραγωγούνται και αυτό φυσικά αυξάνει αυτή την αίσθηση έλλειψης εμπιστοσύνης και κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά και η Guardia di Finanza αλλά και όλοι οι οργανισμοί αντιμετώπισης του φαινομένου αυτό και επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιτυχείς για την ανάκτηση κυρίως των ποσών τα οποία έχουν εκταμιευθεί παρανόμως δεν προβάλλονται αντιστοίχως. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και αυτές οι δράσεις ε, να την χάνουν τις αντίστοιχες προβολής. Και το λέω διότι στο παρελθόν ήμουν εισηγήτρια, εγώ ε, είμαι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μία έκθεση η οποία... Ε, κάνει πολύ στενή σχέση μεταξύ της προβολής αυτού του φαινομένου και του ίδιου του φαινομένου και το πώς ε, το αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη. Και θα ήθελα να προσθέσω και μια δεύτερη πτυχή, ε, κατά την απόψή μου, που αφορά το θέμα της απάτης, που είναι ένα θέμα το οποίο ε, το τελευταίο διάστημα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακούσαμε και από τις παρουσιάσεις εδώ, οδήγησαν και στην ενίσχυση της Όλαφ και τη σύσταση αυτών των ε, εθνικών ε, μονάδων συντονισμού, των ΑΦΚΟΣ και θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση εδώ ε, διότι το ακούσαμε και το αντιλαμβάνομαι και εγώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην άλλη επιτροπή που συμμετέχω είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Ε, είναι οι δύο επιτροπές λοιπόν και οι δύο τομείς που βλέπουν να γιγαντώνεται αυτό το φαινόμενο. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τις πιο συχνές ε, περιπτώσεις απάτης ε, που διαπιστώνεται στο συγκεκριμένο τομέα και αν ε, επειδή ακούσαμε να αναφέρεστε και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία σύμπτωση, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, μήπως θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα θετικά στοιχεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές που για, για μας ως Ιταλία μας χαροποιεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ηγετική θέση, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει σίγουρα να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε όμορφη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, ε, γιατί ε, έτσι θα έχουμε και τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κιέζα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, διότι ούτως ή από τις ερωτήσεις φαίνεται ότι όλοι για τα ίδια ενδιαφερόμαστε. Να συνεχίσω από το, αυτό που ρώτησε η Πρόεδρος Γκρέσλε στην αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, την Guardia Αντιφινάντσα και τους δύο στρατηγούς εδώ για τα όσα κάνουν και Αυτά τα βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβάλλονται και είναι πολύ σημαντικό. Ίσως η ιστορία, όπως είπε και ο στρατηγός Τόσκι, μας οδηγεί να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατία είχαμε ζωφερά χρόνια. Εγώ ήμουν νέο τότε, οι ερυθρές ταξιαρχίες, ε, φαινόμενα της ε, μαφίας που διαρθρώθηκαν σε κάθε ε, διαφορετική περιοχή, οδήγησαν σε ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου της Guardian Finanza τα τελευταία χρόνια. Να συνεχίσω λοιπόν από την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλεφ. Θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τα όσα κάνουμε εμείς στην Ιταλία με το έργο των άλλων χωρών και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει όλα ε, σε αυτό. Αν θυμάστε κυρία Πρόεδρε αναφερθήκαμε στους ε, διαφορετικούς ρόλους πριν από 13-14 χρόνια θα πρέπει ίσως εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα άλμα ποιότητας. Αν μπορείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε, αλλά αν μπορείτε να μας κάνετε κάποια πρόταση. Διότι πραγματικά αυτή η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί, να μπορέσουμε να έχουμε κάτι το οποίο να μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Όλαφ σε όλη αυτή τη δουλειά. Τι μπορεί να κάνει η Όλαφ και τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, καταφέρει ε, διότι τα στοιχεία εδώ είναι εντυπωσιακά. 75% είναι ανησυχητικό στοιχείο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Όλαφ. Πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πιο αποτελεσματική και την Όλαφ. Αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Κλείνοντας ο Πρόεδρος Αχτσουή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι πραγματικά δηλώνω εντυπωσιασμένος ε, από τις παρουσιάσεις σας. Εδώ πρόκειται για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο ενδιαφέρει και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Είναι ένα ζήτημα διακυβέρνησης. Πράγματι, υπάρχει πολυμορφία στην Ευρώπη, δεν έχουμε τις ίδιες μεθόδους σε όλα τα κράτη-μέλη, ούτε καν την ίδια γλώσσα πολλές φορές. Παρότι μιλούμε για ένα έλλειμμα 3% παντού, όμως υπάρχει ένα ε, τεράστιο χάσμα σε ό,τι αφορά την ομοιογένεια και μια τεράστια προσπάθεια που απαιτείται και σε ό,τι αφορά την ε, απάτη και την ε, φόρο αποφυγή. Θεωρώ ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μόνο τα κράτη δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ε, εκτελούν αυτό το ελεγκτικό έργο. Ε, τώρα έχουμε διαφορετικές μεθόδους, ε, τα επίπεδα αποτελεσματικότητας ε, διαφέρουν, άλλες χώρες έχουν πολύ αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου, άλλες όχι. Πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση. Εμείς ε, προσπαθούμε να καταρτήσουμε κανονισμούς ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Και τελικά έχουμε κανόνες σχεδόν ε, αφόρητους. Κανονισμούς μάλλον. Ε, με νομικές βάσεις που και οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι φορείς της αγοράς έχουν τελικά μια σχεδόν ε, εικόνα καρικατούρας ε, της Ευρώπης. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με εσωτερικούς μηχανισμούς όπως αυτούς που ανέπτυξε η Ιταλία. Δεν μπορούμε παντού να εφαρμόζουμε κοινού ε, κανόνες. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Έχουμε χώρες πεντάστερες εντός αγωγικών όπως η Ιταλία και άλλες που υπολείπονται. Και τελικά δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε κι εσείς, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός ε, με όλες αυτές ε, τις ε, συγκεκριμένες λεπτομέρειες και διατάξεις δεν επιφέρει κάτι επιπρόσθετο σε σχέση με αυτούς τους ελέγχους που κάνετε στην Ιταλία. Το δεύτερο ερώτημά μου, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τις υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου και οικονομικής λογοδοσίας. Εσείς είστε αστυνομική υπηρεσία. Ε, οπότε εσείς λογοδοτείτε στη δικαιοσύνη. Μετά, για την Όλαφ. Στον τραπεζικό κλάδο έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουμε και μία ε, αρχή ελέγχου, δηλαδή της ε, τραπεζικές αρχές στις επιμέρους ε, κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης. Ίσως και εδώ να πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες και να υπάρχουν ε, μειονεκτήματα. Όμως ε, η Όλαφ μπορεί να έχει ακριβώς το, το ίδιο εύρος εξουσιών και λειτουργιών σε σχέση με τις εθνικές αρχές και η Όλαφ θα μπορούσε εδώ Ε, να μπορεί να κάνει rating, δηλαδή να βαθμολογεί ε, την ποιότητα των ελέγχων που εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να βοηθούμε και τις ε, εθνικές αρχές. Ε, προκειμένου λοιπόν να μην έχουμε όλους αυτούς τους υπερβολικά λεπτομερείς ε, κανονισμούς ε, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε όλα τα κρατημέλη ακόμα και σε αυτά που έχουν ένα πολύ καλό τρόπο λειτουργίας και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει πράγματι ένα περιθώριο βελτίωσης. Σας ευχαριστώ πάντως και σας συγχαίρω για το έργο σας. Cercherò di rispondere θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά πολλές ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα τα πω λίγο ατάκτος, ελπίζω όμως να είμαι πλήρης. Καταρχάς θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα της κατάρτισης και θα ήθελα να επιστρέψω κυρίως με μεγάλη ευχαρίστηση και με περηφάνεια διότι στις 21 Νοεμβρίου θα γενιέσουμε το έτος ε, μελέτης ε, όλων των ε, Ινστιτούτων Κατάρτισης της Guardia di Finanza και το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για όλη την επόμενη χρονιά και εδώ έχουμε και ένα ιστορικό ημερολόγιο που είναι και ε, ε, πολύ σημαντικό, κυρίως ασχολούμαστε με την κατάρτιση. Πώς η Guardia di Finanza ασχολήθηκε με την κατάρτιση, συνέσβαλε στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της και έδωσε ε, προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Η δέσμευσή μας σε θέματα κατάρτισης αναγνωρίστηκε και το 2014 Το 2017 ανανεώθηκε το πρωτόκολλο συνεννόησης με τον ΩΣΑ ε, για την κατάρτιση στην ε, Σχολή Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Αστυνομίας ε, και ε, διαφόρων τμήματων και μονάδων της αστυνομίας για να μπορέσουν να ε, εξοικειωθούν με τις διαδικασίες της έρευνας ε, σε επίπεδο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ώστε να καταρτιστούν όλοι πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τις διαδικασίες έρευνας διότι πρέπει να μπορούν να μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Να μπορούν λοιπόν να δραστηριοποιούνται όλες οι αστυνομικές δυνάμεις με τον ίδιο τρόπο και αυτό σίγουρα θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα επιτρέψει να έχουμε αποτελέσματα και να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε και να ε, ε, διαλευκάνουμε υποθέσεις απάτης πολύ πιο γρήγορα. Και θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε. Ο παρόν πρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας, ο πρόεδρος Γκράσο, ο οποίος ήταν εθνικός εισαγγελέας καταπολέμησης της μαφίας, ήταν αυτός ο οποίος το 2010-2011 μετέβη προσωπικά στη Σερβία και έγραψε την νομοθεσία κατά πολέμησης μαφίας της Σερβίας βάση της δικής μας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο παρόν πρόεδρος της Γερουσίας λοιπόν ε, ήταν ο πλέον ειδήμων, διότι ήταν εισαγγελέα στη Σικελία, δικαστή συγγνώμη, στη Σικελία για πάρα πολλά χρόνια και ήταν και ειδικό εισαγγελέα για την καταπολέμηση τη μαφία και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Με τη Σερβία έχουμε εντατικότατε σχέσει. Ε, έχουμε επαφές κάθε εβδομάδα και κυρίως από αυτή τη χώρα φίλοι Έχουμε και στην Πρεσβεία έναν επιρογνώμονα για συνεργασία σε θέματα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής απάτης και παρέχουμε στη χώρα αυτή, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, συνδρομή η οποία ε, με... Ε, μαθήματα κατάρτισης ε, για να εκπαιδευτούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταπολεμήσουν την ε, γενικότερη φορολογική απάτη με κυρία αναφορά όμως ε, στην φορολογική απάτη η οποία εμφανίζεται πιο συχνά. Για παράδειγμα, πρόσφατα στο Τριέστε, στην Τεργέστη, είχαμε συνάντηση των Βαλκανικών χωρών πριν από 15-20 μέρες και εκεί συναντηθήκαμε με όλους τους υπουργούς εσωτερικών, όλους τους επικεφαλείς ε, αρχηγούς αστυνομίας των Βαλκανικών χωρών και όλοι μου ζήτησαν να ε, τους φιλοξενήσουμε ε, στο αρχηγείο μας ή στην ε, σχολή της Guardia di Finanza για να οργανώσουμε κύκλους μαθημάτων για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό της αστυνομίας, τους αστυνομικούς των διαφόρων χωρών, Μαυροβούνιο, Αλβανία και αρκετές άλλες, για να μπορέσουν να ακολουθήσουν διαδικασία έρευνας και να μπορέσουμε να έχουμε μια εναρμόνιση της νομοθεσίας. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και το βουλευτή που ε, επένεσε την Guardia di Finanza και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εκείνους που αναγνώρισαν ότι η Guardia di Finanza επιδεικνύει ιδιαίτερο επαγγελματισμό. Επαγγελματικός ο οποίος απορρέει από πάρα πολλά χρόνια ε, καταπολέμησης οργανώσεων της μαφίας, τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά κυρίως εγώ θα έλεγα γιατί η Ιταλία είναι μία από τις λίγες χώρες ε, ε, διότι ε, όλες οι χώρες του κόσμου θα θέλαμε να έχουν ε, ένα τμήμα της αστυνομίας που να είναι σαν την Guardia di Finanza. Είναι ελάχιστες οι χώρες, δεν λέω κανείς, δεν λέω ότι είναι μοναδική η Guardia di Finanza από καταπόλυτο τρόπο, αλλά ε, σίγουρα δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες ε, δομές όπως η Guardia di Finanza. Δηλαδή ένα σώμα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστυνομίας, ε, της οποίας η αστυνομική πέραν ε, των καθηκόντων της δικαστικής αστυνομίας είναι και φορολογική αστυνομία, ε, αστυνομία που αφορούν και την ε, δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια σε κάποιες περιπτώσεις. Συνεργάζονται λοιπόν και για την δημόσια τάξη σε κάποιες περιπτώσεις, αν και πάντα με γνώμονα την οικονομική και χρηματοπιστωτική απάτη. Κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω σίγουρα, αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα τα ανέφερα και για τα οποία είμαστε πολύ περηφανοί και σας παρουσιάσαμε εδώ σήμερα με κάποια περηφάνεια, αλλά και εμείς ανησυχούμε ε, για τα αποτελέσματα. Γιατί, διότι προφανώς η απάτη, παρά το γεγονός ότι βελτιώνει την νομοθεσία και η κινητική νομοθεσία ε, πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ε, απάτης. Και γι' αυτό ακριβώς ε, η Guardia di Finanza, και εδώ έρχομαι να απαντήσω και σε μια περαιτέρω ερώτηση, επειδή ακριβώς είναι οικονομική και χρηματοπιστωτική αστυνομία και αυτή είναι η ερώτηση μου έθεσε η κυρία Κινίτσι, η σχέση με τις φορολογικές υπηρεσίες, την Επιτροπή Οικονομικής Χρηματοπιστωτικής Ασφάλειας που σύστησε ο Υπουργός ε, Οικονομικών και Οικονομίας καθορίστηκε ότι οι συνάδελφοι ε, των ε, φορολογικών διοικήσεων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της φορολογίας. Δηλαδή, τη διαχείριση του κάθε φορολογουμένου από τη στιγμή που αποκτά αριθμό φορολογικού μητρώου μέχρι ε, το τέλος ε, του δίνεται φορολογική βοήθεια, ε, παρακολουθείται ε, η, διαδικασία της ε, φορολογίας κλπ. Η Guardia di Finanza είχε πάντα ευθύνη αντιμετώπισης και καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και κυρίως ε, ε, υπήρχε και το διεθνές στοιχείο και εδώ απαντώ και σε ε, περαιτέρω ερώτηση τις απάτες τύπου καρουσέλ η απάτη τύπου καρουσέλ είναι κλασική έκφραση θα έλεγα σχολικού τύπου ε, της απάτης που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται δηλαδή από μη καταβολή φόρων σε διεθνές επίπεδο ε, και αυτό προκαλεί μεγάλες ε, ζημίες, ε, όχι μόνο σε οικονομικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχει και μια πτυχή που εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ και μας απασχολεί και πάρα πολύ, του ανταγωνισμού. Διότι το θέμα του ανταγωνισμού, η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη, οποιαδήποτε παρανομία σε φορολογικό επίπεδο δεν δημιουργεί μόνο οικονομικές ζημίες, αλλά δημιουργεί και μια μεγάλη στρέβλωση στους ε, κανόνες του θεμητού ανταγωνισμού. Και έτσι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει, αυτός ο οποίος ε, δεν θέλει να καταβάλει τους φόρους του ή επιλέγει να μην καταβάλει τους φόρους του, ε, μπορεί να έχει κάποια κέρδη τα οποία στην καλύτερη περίπτωση ισοδυναμούν με μη καταβολή ΦΠΑ Επομένως, ε, σε εμπορικό επίπεδο δεν καταβάλει ένα 20%. Ένα 20% σε εμπορικό επίπεδο σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στρέβλωση ε, του ανταγωνισμού. Θα προσπαθήσω να απαντήσω επίσης ε, και στην ερώτηση που έγινε όσον αφορά τις τράπεζες και τα τραπεζικά ιδρύματα. Επιτρέψτε μου εδώ και πάλι με μεγάλη περηφάνεια να διεκδικήσω το ιταλικό στοιχείο από το 1976 με το νόμο 159 του 1976, δηλαδή την εισαγωγή της λεγόμενης νομοθεσίας ε, αξιολόγησης, Για τα μέλη της Guardia di Finanza υπάρχει μια συγκεκριμένη μονάδα που από το 1976 χέρι των ίδιων εξουσιών ε, πρόσβασης, επιβεβαίωσης και επομένω ελέγχου που ήδη αναγνωρίζονταν στους ε, ε, υπαλλήλους της Τράπεζας της Ιταλίας. Από το 1976 πρόκειται για μια ειδική μονάδα που στην αρχή ήταν ένας περιορισμένος αριθμός στρατιωτικών, αλλά τώρα πια είναι πολύ περισσότερα μέλη της Guardia di Finanza. Υπάρχει ο νόμος 413 ε, ο οποίος αφορά κυρίως ε, τους τραπεζικούς ελέγχους στα πλαίσια ε, οικονομικών ερευνών και γίνεται δυνατό, υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να μπορέσει κάποιος να ελέγξει την τραπεζική κατάσταση, τους λογαριασμούς δηλαδή κάποιων υπόπτων για φοροδιαφυγή, για φορολογική απάτη και πέραν αυτού και οικονομικών εγκλημάτων. Γίνεται παντού αυτό, με ρωτάτε. Είναι τόσο εύκολο να γίνονται αυτές οι έρευνες ε, σε διεθνές επίπεδο. Η απάντησή μου εδώ είναι ότι δυστυχώς όχι. Ε, δεν ισχύει παντού το ίδιο. Δεν ε, βρίσκουμε σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στις ε, βόρειες χώρες της Ευρώπης, την ίδια νομοθεσία, τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης και συνεργασίας και την ίδια δυνατότητα ε, συντονισμού. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς θα συνεχίσουμε και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά, όχι μόνο ε, μέσω διεθνών σχέσεων που έχουμε, αλλά προσπαθούμε και να δημιουργήσουμε και πιο αυστηρές μορφές συνεργασίας, όχι μόνο σε δικαστικό επίπεδο, ε, εδώ νομίζω ότι θα προσθέσει και κάτι ή θα μπορούσε να προσθέσει κάτι ο Υπουργός, αλλά ε, σε διοικητικό επίπεδο. Και με αυτό ολοκληρώνω και ζητώ συγγνώμη αν ε, μακρηγόρησα. θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την κοινή κατάρτιση που θεωρώ ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε όλοι καλύτερα και να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε όλοι την ίδια επιχειρησιακή γλώσσα, ας το θέσω έτσι, και επομένως να προσπαθήσουμε να ε, επιταχύνουμε και να μειώσουμε και τις ε, διαδικασίες και ε, ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να βοηθούμε σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο κατάρτισης αλλά σε και επίπεδο ενεργού συνεργασίας ε, ε, με τις δικαστικές αρχές. Τι πόρους διαθέτεται. Τι πόρους διαθέτεται. Χρήματα. Η Guardia di Finanza αυτή τη στιγμή αριθμεί 58.000 άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει όμως ε, μία πρόβλεψη για αναδιάρθρωση όλων των αστυνομικών ε, δυνάμεων, ο λεγόμενος ε, νόμος Μαντία, ο οποίος εγκρίθηκε φέτος και επομένως θα γίνουμε περίπου 63.000. Θα έχουμε δηλαδή 63.000 μέλη. Πρόκειται για έναν αριθμό ο οποίος ε, πρόσφατα από μια εξέταση που έκανε η κυβέρνησή μας θεωρείται ότι αρκεί, ελπίζω να αρκεί γιατί τα καθήκοντά μας είναι πολλά, η δέσμευση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά ε, και στο μέλλον. Ναι, πολύ σύντομα κι εγώ, γιατί νομίζω ότι ο στρατηγός ε, Τόσκι απάντησε ε, πλήρως στις ερωτήσεις. Ήθελα όμως ε, να κάνω δύο παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της καταπολέμησης της απάτης είναι ένας τομέας ε, ιδιαίτερα σημαντικός ε, της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για δύο λόγους. Καταρχάς, ε, διότι προστατεύουμε την οικονομική ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κανόνες, νόμος, να εφαρμόζονται σωστά όλα όσα προβλέπονται σε κοινοτικό επίπεδο. Και το δεύτερο, γιατί από πολλές σκοπιές και νομίζω ότι εδώ έρχομαι να συμφωνήσω με αυτά που έλεγε ο κύριος ε, Αρτουή, η κυρία Κινίτση και ο κύριος Τσέζε. Υπάρχει και ε, πολύ μεγάλη ε, σημασία επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς πολιτών. Χρειάζονται σίγουρα εθνικές αρχές οι οποίες θα έχουν τα κατάλληλα και η μήτρα θα είναι κατάλληλα οργανωμένες και θα έχουν και την κατάλληλη δέσμευση. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη αυτές οι εθνικές αρχές ε, να συνομιλούν, να συνεργάζονται αλλά υπάρχει και ένα όριο πέραν του οποίου η οριζόντια συνεργασία μεταξύ των αρχών δεν μπορεί να φτάσει πρέπει να υπάρχει ε, και μία ε, κάθετη, αν θέλετε, διάσταση σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει λοιπόν το θέμα των κοινών προτύπων. Πρέπει κάποιος να τα καθορίσει αυτά τα κοινά πρότυπα. Και ο οριζόντος διάλογος δεν αρκεί για να καθορίσουμε κοινά πρότυπα. Και εδώ έρχομαι να συμφωνήσω με αυτό που είπε προηγουμένως ο στρατηγός Ατάρτη και ο στρατηγός Τόσκι. Και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος θα αποτελεί ένα κόμβο συντονισμού ή ε, ε, ίσως και κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι ένας από τους τομείς όπου ίσως αυτό το κάτι παραπάνω χρειάζεται. Η Ιταλία σίγουρα έχει κάνει συγκεκριμένη επιλογή ε, να αναπτύξει περαιτέρω τις ε, δυνατότητες που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι τυχαίο ότι εμείς έχουμε προτείνει την ενισχυμένη συνεργασία για να υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ού μόνον αυτό, επιμείναμε και με τους εταίρους μας, διότι θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ περιορισμένες οι αρχικές αρμοδιότητες που θέλαμε να αναθίσουμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είπαμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να χρησιμεύσει και σε άλλους τομείς. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για παράδειγμα, είναι ένας άλλος τομέας, στον οποίο η οριζόντια συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών όσο επαγγελματίες και να είναι, όσο ικανοί και ε, κατάλληλα οργανωμένοι να είναι, δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει και διασυνοριακή αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων. Και η Ιταλία έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή, αλλά πρέπει να σας πω ότι τρόπον την Α, ε, όπως ε, πολύ σαφώς παρουσιάστηκε σήμερα, και η Guardia di Finanza και σε γενικά έσγραμμες οι Ιταλικές αρχές έκαναν μια πολύ σαφή επιλογή και θα το πω με ε, κάτι αγγλικό, με έναν αγγλικό όρο. Engage η Guardia di Finanza απέδειξε ότι δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει ζήλια μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων της τάξης. Ε, απλώς αποδυναμώνει τη θέση τους. Η Ιταλία απέδειξε ότι δεν χρειάζεται ε, να υπάρχει engagement μόνο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους άλλους εταίρους. Πρέπει να το αναζητήσουμε, πρέπει να το παντρευτούμε αυτό το engagement. Και αυτό ε, αποδεικνύει ότι αυτή η στάση ε, η τάση να συνεργαζόμαστε, να διαθέτουμε πόρους και να είμαστε και διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και να κάνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια ε, μπορεί να ξεκινήσει και να δράσει ως πολλαπλασιαστικός παραγόν για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα από ένα σώμα όπως είναι η Guardia di Finanza. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προσθέσω ε, ένα πολύ μικρό στατιστικό στοιχείο στα όσα είπε ο διοικητής και να απαντήσω λίγο και στον κύριο Τσεχόφσκι. Το συγκεκριμένο στοιχείο αφορά τη διαφοροποίηση τρόπων ε, λειτουργίας που υπάρχουν, ε, τρόπων modus operandi. Είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου να το πούμε αυτό. Στον τομέα των ελέγχων, στον τομέα των δαπανών, έξι χώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο έξι χώρες επιτρέπουν ε, να μπορεί κάποιος να πάει να κάνει έλεγχο στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Σε 11 χώρες πάντα χρειάζεται δικαστικό ένταλμα και μάλιστα σε πέντε χώρες δεν μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση. Άλλη πτυχή. Μόνο σε πέντε χώρες μέλη μπορεί κάποιος να κάνει χωρίς περαιτέρω έγκριση ε, διαδικασίες σήμανσης ε, και ε, δέσμευσης υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων κλπ. Σε εννιά χρόνες, χώρες μπορεί να γίνει μόνο μέσω δικαστικού εντάλματος και σε άλλες εννέα χώρες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Από αυτό και μόνο ε, φαίνεται σαφέστατα τι διαφορά υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό κατά συνέπεια. Και επιτρέψτε μου εδώ για να ε, συνεχίσω να μιλάω για αυτό το ιταλικό στοιχείο. Η Ιταλία ε, δεν είναι το μαύρο πρόβατο το οποίο ε, μα θεωρούσαν τόσα χρόνια. Από πού προέκυπτε αυτό το μαύρο πρόβλητο. Το γεγονό ότι στην Ιταλία είχαμε αυξημένο αριθμό περιπτώσεων, το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχαν περισσότερε παρατυπίες στη συγκεκριμένη χώρα. Στην πραγματικότητα υπήρχε απλώς μεγαλύτερος έλεγχος. Έλεγχος ε, ο οποίος γινόταν ε, επειδή υπήρχαν μεγαλύτεροι, περισσότεροι λογιστικοί έλεγχοι, πιο καλά εκπαιδευμένοι και ελεγκτές ε, πιο καλή και αυτό επιτρέπει να διαπιστώνονται πολύ περισσότερες παρατυπίες. Επομένως, οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλό ποσοστό παρατυπιών έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης ε, σε σχέση με χώρες που έχουν χαμηλότερο ποσοστό παρατυπιών. Τώρα, για να απαντήσω στον Τσέχο Ευρωβουλευτή. Συμφωνώ απολύτω με την πρότασή σα. Είναι εξαιρετική ιδέα. Εμείς ως Ιταλία ε, αναφέρθηκα στο νέο ε, πρόγραμμα συνεργασίας. Ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει είναι ακριβώς να διευρύνουμε ένα σχέδιο συνεργασίας ε, με κατάρτιση κοινή, κοινή εκπαίδευση μέσω της άμεσης ε, ε γνώσης μέσω των ΑΦΚΟΣ και το ΑΦΚΟΣ της Τσεχίας είναι αυτό το οποίο απάντησε ταχύτατα και συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Αυτή η ανταλλαγή λοιπόν σίγουρα θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια. Αυτά ήθελα λοιπόν μόνο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, στρατηγία, έχετε κάνει μία αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε μία από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε αν ότι ε, κάποιες χώρες επιτρέπουν ε, την πρόσβαση ε, στους εμπορευόμενους και άλλες όχι θα μπορούσατε να μας ε, δώσετε αυτή την αξιολόγηση αναχώρα για να ξέρουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση της Ένωσης. Αν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να το αναφέρουμε, όχι μόνο να μιλούμε για γενικά στατιστικά στοιχεία και ε, να υπάρχουν και οι απαραίτητες επιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να κλείσω τώρα τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τι διερμηνέ που μα έδωσαν λίγο παραπάνω χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ομιλητέ μα σήμερα εδώ για την προσέλευσή του και τι ε, πληροφορίε που μοιράστηκαν ε, μαζί μα, σημαντικέ πληροφορίε και φυσικά το δικό μα to-do list είναι μεγαλύτερο από το δικό σα, αλλά τα όσα μα είπατε εδώ πραγματικά μα δώσαν ε, πολύ τροφή για σκέψη. Σα ευχαριστώ και πάλι θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ και μάθαμε πολλά σήμερα από εσά. Σα ευχαριστώ πολύ.